Friends, this αρχίσουμε λοιπόν, θα έρθουν και οι υπόλοιποι, έχουμε ε, μετάφραση σε όλες τις ε, γλώσσες με εξαίρεση τα κροατικά. Επιθυμώ επίσης να σας πω ότι έχουμε και ομάδες επισκεπτών της κυρίας Μωράν Σατιέ ομάδα 10 δημοσιογράφων, για να παρακολουθήσουν την ψηφοφορία της εκθέσεως για τους αποσπασμένους εργαζομένους και ορισμένοι θα βιντεογραφήσουν και τμήματα της ε, ψηφοφορίας και ο κύριος Σούλτσε έχει προσκαλέσει μια ομάδα ε, μαγνητοσκοπητών που θα ε, μαγνητοσκοπήσουν επίσης και ο κύριος Σιλικιώτης, όταν θα έρθει βέβαια, θα υποδεχθεί ομάδα 55 επισκεπτών για το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, δηλαδή την κοινή ακρόαση Εμπλτραν. Αναμένουμε την κυρία Ντελή για να προσέλθει. Νομίζω πάντως ότι, χωρίς να φανούμε βεβαίω αγενείς, αλλά για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε καθώς ε, η κυρία Ντελή θα καταφθάνει, θα αρχίσουμε την ακρόαση για τις ε, συνθήκες εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων στις μεταφορές. Των μετακινούμενων εργαζομένων στις μεταφορές. Απευθύνω το καλώς ορίσατε σε όλους τους επισκέπτες και ιδίως τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη τους μαζί μας. Ε, μας ικανοποιεί πολύ που συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Μεταφορών και ως γνωρίζετε οι οδικές μεταφορές είναι και ο πιο κύριος τρόπος μεταφορών. Το 2014 τα τρία τέταρτα περίπου, τρία τέταρτα όλων των εσωτερικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασαν από τον δρόμο. Και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επιβατών, οι ε, οδικές μεταφορές αφορούν το άνω των 90% όλων των επιβατών. Καλώς ήρθατε κυρία Ντελή. Άρχισα με μια σύντομη εισαγωγή κυρία ε, Ντελή για να μην χάσουμε χρόνο γιατί μετά έχουμε και ψηφοφορία. 10,6 εκατομμύρια πρόσωπα εργάζονται στον τομέα μεταφορών, 10,6 εκατομμύρια επαναλαμβάνω, δηλαδή πολλοί άνθρωποι. Και η αξιολόγηση έχει δείξει ότι η κατάχρηση των κοινωνικών κανόνων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση επισύρουν σημαντικά προβλήματα με ε, ιδιαίτερα επιβαρημένα ωράρια εργασίας των επαγγελματιών οδηγών σε σχέση με άλλους τομείς επαγγελμάτων, με άλλους επαγγελματίες. Υπάρχουν και ε, σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, ε, για παράδειγμα μακρά διαμονή μακριά από τις αιστείες τους, ανεπαρκείς εγκαταστάσεις ε, παραμονή του και άλλα. Αυξάνουν αυτά τα πράγματα το κόστος του ανταγωνισμού και οδηγούν σε παράνομες πρακτικές που διευρύνουν το πρόβλημα. Και τα υψηλά κόστη όχι μόνο στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, αλλά οδηγούν και στον κίνδυνο στέρησης των οδηγών από τα δικαιώματά τους, όταν εργάζονται προσωρινά σε άλλες χώρες μέλη, διότι υπάρχουν υψηλότερα κίνητρα για τις άλλες επιχειρήσεις για να καταστρατηγούν τους κανόνες. Λόγω του χαρακτήρα του επαγγέλματος αυτού χρειάζεται ειδική νομοθεσία για τον τομέα αυτό που κρίνεται ότι είναι η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. και λαμβάνονται και άλλες πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσουν την κατάσταση στην εσωτερική αγορά μεταφορών. Στη... Τον Μάιο ήδη φέτος με το πλαίσιο Europe on the Move η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την ε, απόσπαση των ε, οδηγών με πρόταση για ελάχιστες απαιτήσει για τις περιόδους αναπαύσεως, για τους ταχογράφους και την πρόταση για την ε, πρόσβαση στις σχετικές αγορές. Σήμερα η σημερινή ακρόαση θα τροφοδοτήσει την συζήτηση που διεξάγεται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την συζήτηση αυτή και θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα την ε, συνάδελφό μου, συμπρόεδρο και εμπειρογνώμονα σε θέματα μεταφορών, κυρία Ντελή, να... που είναι επικεφαλής της ε, Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού, να προβεί σε σχετική εισαγωγή. Κυρία Πρόεδρε, Είναι μεγάλη η χαρά για μένα που μπορώ να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ. Σήμερα η αγορά ε, των ε, μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων έχει κρίσιμη σημασία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το όραμα που έχουμε και που ε, προσπαθούμε να μεταφέρουμε είναι ένα όραμα ενός τομέα που θα χρειαστεί αύριο να είναι στέρεος, ε, βιώσιμος, αλλά και σταθερός, ο οποίος θα προσφέρει την δυνατότητα ασφαλώς για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά, αλλά ιδίως να είναι σταθερός ο τομέας αυτός, ώστε να οδηγήσει σε ισότητα μεταχείρισης όλων των Ευρωπαίων εργαζομένων με ένα χρυσό κανόνα που θα πρέπει να είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταφέρει ψηλά το λάβαρο της εργασίας, ε, της ισότιμης μεταχείρισης των εργαζομένων. Να είναι καλές οι συνθήκες εργασίας των ε, προσώπων αυτών. Όπως ακούσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει νέα νομοθεσία για τις χερσαίες μεταφορές, οδικές μεταφορές οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία αυτή όντως θα βελτιώσει την εργασία των εργαζομένων του τομέα και να στηρίξει όλους εκείνους που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν στον τομέα αυτό, ώστε να σέβονται τους ισχυώδεις κανόνες. Συνεπώς, τα θέματα αγοράς και τα κοινωνικά θέματα θα αντιμετωπιστούν από κοινού για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και των συμφερόντων των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πει σημαντικό ρόλο. Η, η συμβολή του θα είναι σημαντική στο θέμα αυτό για να γίνουν σεβαστοί οι στόχοι του και να επιτευχθούν. Για να γίνει αυτό, οφείλουμε να ρυθμίσουμε με κοινή προσπάθεια το ζήτημα του κοινωνικού dumping, που είναι αυτό που δηλητηριάζει το ευρωπαϊκό ε, όραμα. Αναμένω συζήτηση με τις συνεισφορές όλων, αλλά συνεισφορές συγκεκριμένες που να μας επιτρέψουν πραγματικά να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, αλλά και να λύσουμε όλα τα προβλήματα που βλέπουμε καθημερινά στις χώρες μας. Αληθεύει ότι στην συζήτηση που θα διεξαχθεί σήμερα η συζήτηση μάλλον που θα κάνουμε σήμερα είναι μια σημαντική συμβολή αλλά δεν πρέπει να κρύβουμε το πρόσωπό μας απέναντι στα πραγματικά προβλήματα που είναι το πρόβλημα του ελέγχου των ε, εικονικών επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων επίσης, των ζητημάτων επίσης, ας πω καλύτερα, που δεν αναφέρονται μονάχα στον ελάχιστο μισθό, αλλά και στις συνθήκες, είτε πρόκειται του καταλήμματος, είτε των ε, ίδιων των συνθήκων των μεταφορών. Και εν πάση περιπτώσει, κυρία Πρόεδρε, υπενθυμίζω, επαναλαμβάνω, ότι η δική σας επιτροπή, όπως και η δική μου, έχουν ένα μοναδικό στόχο. Να στηρίξουμε, να υπερασπιστούμε το σύνολο των Ευρωπαίων εργαζομένων. Στα συμπεράσματα της εκθέσεώς μας δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Θέλουμε οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια προστασία. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και πάντως μπορείτε να στηρίζεστε στην αποφασιστικότητα των μελών της Επιτροπής Μεταφορών που ήδη είναι πολυάριθμα μέσα στην αίθουσα για την συμμετοχή τους στην ε, συζήτηση. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος κυρία Ουλφσκογκ, κυρία Πρόεδρε Ντελή, για τα εισαγωγικά σας λόγια. Έχουμε τώρα πέντε εμπειρογνώμονες που έχουμε προσκαλέσει και θα ήθελα να τους ακούσουμε. Η κυρία Βαντεπέλτ πρώτα θα ακολουθήσει ο κύριος Ρομπέρτο Παρίλο, ο κύριος Βρόνσκι, ο κύριος Έγκελχαρτ και ο κύριος Ροδρίγε Μεντάλ. Όμως θα αρχίσουμε με την κυρία Βαντεπέλτ που είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ε, Οδικών Μεταφορών. Θα σας διακόψω όμως αν ε, μακρηγορήσετε. Η κυρία Βάντερ Πέλτ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να είμαστε σήμερα εδώ και να δώσουμε τη γνώμη μας σε σχέση με την οδηγία για τις οδικές μεταφορές και τους μετακινούμενους εργαζόμενους, ε, τους αποσπασμένους. Καταρχάς, θα πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστε αμοιβέ και οι κανόνες περί ε, αμοιβόμενη άδεια όταν οι οδηγοί κινούνται στους δρόμους των κρατών μελών. Ε, σήμερα προβλέπεται ότι η η πρόταση λέει ότι όταν μία μετακίνηση είναι πάνω από τρεις μέρες σε κάποιο ε, κράτος μέλος υποδοχής, τότε σημαίνει ότι είναι αποσπασμένο αυτό το κράτος και άρα μετρών ε, η μήνυμο αμοιβή και οι ε, οδηγίες περί ε, αμοιβόμενων διακοπών. Όταν όμως η διαδρομή είναι λιγότερη από τρεις μέρες, μάλλον είναι ίση με τρεις μέρες, τότε σημαίνει πως δεν είναι αποσπασμένος και ότι ισχύουν τα περί καμποτάζ. Αυτό που είναι νέο είναι πως η πρόταση περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες για τη μέτρηση του τριήμερου αυτού λέει πως μια ημερήσια εργασιακή διάρκεια έξι ωρών είναι μισή μέρα, ενώ όταν είναι πάνω από 6 ώρες είναι ολόκληρη, θεωρείται ολόκληρη μέρα. Επίσης όταν έχει ανάπαυση, διάλειμμα ή έχει, είναι σε διαθεσιμότητα στην επικράτεια του κράτους ή μέλους υποδοχής, αυτές οι περίοδοι θεωρούνται περίοδοι εργασίας και άρα καταμετρώνται για να μετρηθεί αν είναι απόσπαση ή όχι. Όσον αφορά την ξεκάθαρο ορισμό της ίδιας της απόσπασης υπάρχουν κάποιες σημαντικές ελλείψεις. Ας πούμε όταν, είναι, όταν ε, υπάρχει διέλευση. Πουθενά δεν αναφέρεται η διέλευση στην πρόταση. Εμείς πιστεύουμε πως θα πρέπει ρητά να αναφέρεται γιατί η διέλευση ποτέ δεν θεωρείται ως απόσπαση και υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες όσον αφορά τον, τον όρο μήνυμου αμοιβή. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ε, επιδόματα ημερήσιας αποζημίωσης ή οποιασδήποτε είδος αποζημίωσης, ε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας ξεχωριστός σύνολο κανόνων. Θα ήταν καλύτερο να ορίσουμε τι θεωρείται ελάχιστη αμοιβή και τι όχι να υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος δηλαδή στοιχείων που θεωρούνται μετρώμενα μέσα στην μήνυμη αμοιβή, γιατί αν δεν υπάρχει σαφής ορισμός, η συζήτηση για το κατά πόσο τηρείται η μήνυμη αμοιβή θα ε, συνεχιστεί. Εν γέννη θεωρούμε πως είναι πολύ θετικό που επιτέλους έχουμε σαφή ορισμό του τι θεωρείται απόσπαση και τι όχι, καθώς και σαφείς ε, κανόνες υπολογισμού. Ωστόσο φοβόμαστε πως η ο προτινόμενος κανόνας των τριών ημερών θα είναι μειονέκτημα για τα μικρομεσαίες και τα μικρά και επίσης για τις εταιρείε που ε, έχουν έδρα στα περιφερειακά κράτη-μέλη. Ένα παράδειγμα μπορεί να αποσαφηνίσει αυτή μας την άποψη. Ένα παράδειγμα, αν πάρουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση που φεύγει από την Ισπανία και μεταφέρει πορτοκάλια από την Ισπανία στις κάτω χώρες. Μια, ένα ε, ταξίδι μιας εβδομάδας μέχρι την Ολλανδία και πίσω. Ο οδηγό ξεκινά από την Ισπανία. Θα διασχίσει την Γαλλία για περίπου δύο μέρε, το Βέλγιο μισή μέρα και θα φτάσει τελικά στι κάτω χώρε όπου θα ξεφορτώσει και θα ξαναφορτώσει το φορτίο επιστροφή του για το Βέλγιο και για τη Γαλλία η διέλευση από τη Γαλλία και το Βέλγιο στην πορεία προς την Ολλανδία είναι διέλευση, άρα δεν θα θεωρηθεί ποτέ ως αποσπασμένος. Θα ξεφορτώσει και θα φορτώσει στην ε, Ολλανδία πάνω από 6 ώρες, οπότε μια ολόκληρη μέρα θα μετρηθεί. Θα επιστρέψει στο Βέλγιο, θα ξεφορτώσει εδώ μέρος του φορτίου επιστροφής, λιγότερο από 6 ώρες θα μείνει εκεί, οπότε θα μετρήσει μισή μέρα στο Βέλγιο, θα συνεχίσει στη Γαλλία και οι δραστηριότητε του εκεί θα του πάρουν πάνω από μία μέρα και έξι ώρες, δηλαδή θα μετρήσει δύο μέρες. Και ο ίδιος οδηγός κάνει αυτή τη διαδρομή 4 με πέντε φορές το μήνα. Επί τη βάση των κανόνων για τον υπολογισμό, ο άνθρωπος αυτός θα είναι αποσπασμένος στη Γαλλία για 10 μέρες περίπου, στην Ολλανδία για περίπου 4 με 5 μέρες και ίσως και στο Βέλιο για 3 μέρες αναλόγως τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του στο Βέλγιο. Και για να καταστεί ακόμη πιο δύσκολο, που και που θα κάνει και λίγο καμποτάζ από Λουξεμβούργο, δηλαδή εκεί θα πρέπει να πληρωθεί αμοιβή Λουξεμβούργου για τις λίγες ώρες που θα περάσει εκεί. Για το ολόκληρο το μήνο του όμως η κοινωνική του ακάλυψη είναι από την Ισπανία. Για να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία ο εργοδότης θα πρέπει να κάνει κάθε μήνα να κάνει περίπλοκους προπολογισμού για κάθε οδηγό του που έχει διαφορετικές διαδρομές να κάνει. Αυτός ο εργοδότης θα πρέπει να γνωρίζει τους μισθούς καθώς και τους κανόνες για τις υπερορίες και για τις αποζημιώσεις αλλά και για τις διακοπές ε, και για την άδεια σε όλες τις χώρες που περνά ο οδηγός. Οι εργοδότες, ε, κυρίως οι μικρομεσαίες, ε, θα πρέπει να προσλάβουν ειδικέ εταιρείε συμβουλευτικές που γνωρίζουν τις διαφορετικές νομοθεσίες στα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί οι μικρομεσαίες συνήθως δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να ελέγξουν και να εφαρμόσουν όλο αυτό, όλους αυτούς τους κανόνες οι ίδιοι. Και κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή, κάθε φορά που ο οδηγός πάει σε νέε χώρε, περνάει από άλλε χώρε, ο εργοδότη θα πρέπει να κάνει νέου υπολογισμού ξανά, μανά, κάθε μήνα. Αυτοί οι κανόνες λοιπόν θα δημιουργήσουν τεράστιο φόρτο για τις εταιρείε και δεν θα είναι ε, ε, εύχρηστοι. Οι νέοι κανόνες επίσης μπορεί να οδηγήσουν σε αβεβαιότητα για τους ε, οδηγούς, γιατί θα υπόκειται σε διαφορετικού και νομοθεσίες κάθε μήνα. Η πρόταση επίσης προβλέπει κάποιους κανόνες για τις ε, διοικητικές υποχρεώσεις. Η UTR βλέπει πως με ευχαρίστηση που δεν χρειάζεται πλέον κάποιος εκπρόσωπος γιατί είναι πολύ αυτό δαπανηρό. Ωστόσο, η πρόταση προβλέπει διάφορες υποχρεώσεις καταγραφής που μπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν επίσης υποχρεώσεις για τον ε, οδηγό ώστε να έχει συγκεκριμένα έγγραφα στο φορτηγό του. Και για μια φορά λοιπόν ε, ακόμα ζητάμε μια νέα πλατφόρμα για την καταχώρηση. Αυτό ενδεχομένω ε, να δίνει και τη δυνατότητα να ανεβάζονται τα απαραίτητα έντυπα, το Α1, η σύμβαση εργασία, ίσω άλλα έγγραφα και έτσι ο εργαζόμενο, ο οδηγό. Δεν χρειάζεται να έχει συνέχεια μαζί του έγγραφα αυτά. Μια τέτοια πλατφόρμα θα απλοποιούσε την ε, διαδικασία για τον ε, εργοδότη και θα διευκόλυνε ασφαλώ και τον ε, οδηγό που δεν θα χρειαζόταν να έχει τα έγγραφα αυτά μέσα στο φορτηγό πλέον. Και έτσι θα περιοριστεί και ο κίνδυνο ασφαλμάτων, να ξεχαστεί κάποιο έγγραφο και το θα θέλαμε να υποδείξουμε και άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το κόστος ε, του αθέμητου ανταγωνισμού. Στην τρέχουσα κατάσταση. Έχουμε τεράστιες διαφορές για το εργασιακό κόστος. Ε. Άλλοι δουλεύουν ε, και πληρώνουν τριπλάσια για την ίδια εργασία που γίνεται σε άλλες χώρες και υπάρχουν και μεγάλες διαφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Άρα θεωρούμε ότι το μέτρο δεν θα αλλάξει στην ουσία το πρόβλημα το οποίο είναι το κόστος εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λάκη Πρόεδρος. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρομπένιο Παρίγιο, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ETF στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών. Έχετε το λόγο, κύριε Παλιό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βουλευτές. Να πω στο ζουμί του θέματος. Δεν θα σας κάνω παρουσίαση με διαφάνειες. Θα προσπαθήσω να σας πω ποια είναι τα ουσιαστικά ζητήματα για μας. Είναι δύσκολο σήμερα να αγνοήσει κανείς τις μεγάλες ουρές των φορτηγών ε, που μπλοκάρουν τους αυτοκινητοδρόμους και αυτό έχει παρατηρηθεί από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το, η πρόσφατη επίσκεψη του ETF ε, στα σημεία σταθμευσής ε, στον Οκτώβριο του 2017 αποκάλυψαν πραγματικά φρικτές συνθήκες εργασία σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες οδηγούς όταν επί εβδομάδες και μήνες ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν μας λέει φυσικά κάτι καινούριο. Οι χώρες δεν έχουν υγειονομική ε, εγκαταστάσεις ε, ε, οι οσμοί των ούρων, ε, ε, οι οδηγοί που ετοιμάζουν τα γεύματά τους μέσα στα φορτηγά και έξω. Και είναι χιλιάδες οι οδηγοί που βρίσκονται και ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Και το ETF λοιπόν έχει ξεκινήσει μια σταθερή και διαδρομένη επαφή με αυτούς μέσω των κοινωνικών μέσων. Και οι πιο πολλοί είναι Ρουμάνοι και Βουλγαροί και, και και οι προτάσεις λοιπόν που έχουν γίνει στα πλαίσια του πακέτου της κινητικότητας θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε τους ε, συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες ζωής, γιατί πραγματικά η εικόνα είναι ζωφερή. Έχουμε και εκπροσώπους του BGL, που, μια οργάνωση που επίσης ασχολείται και με τα απορρίμματα. Και την προηγούμενη εβδομάδα στο Βουκουρέστη συναντηθήκαμε με μια ομάδα οδηγών που εργάζονται για σκανδιναβικέ εταιρείε που κάνουν λοιπόν μεταφορά απορριμμάτων από τι σκανδιναβικέ χώρε προ την Γερμανία κυρίω. Και μας κατέδειξαν, δείξαν φωτογραφίες ε, που συλλέγουν τα απορρίμματα. Και δεν υπάρχει κανένα ε, προστατευτικό εξοπλισμό για να μαζεύουν τα απορρίμματα και ούτε αποζημιώνονται τελικά γι' αυτό οι οδηγοί. Και αν σε περίπτωση που παραπονεθούν, του απολύουν πάρα αυτά. Και είναι πεπισμένοι ότι του μεταχειρίζονται έτσι μόνο και μόνο επειδή είναι Ρουμάνοι και είναι και ευάλωτοι και δεν είναι σε θέση να αντισταθούν και να ζητήσουν την εφαρμογή του νόμου. Και είμαι σχεδόν απόλυτα βέβαιος και πεπισμένος ότι οι ενώσεις οι διάφορες θέλουν να βελτιώσουν τους όρους ε, εργασίας των επαγγελματιών ε, οδηγών. Και οι κοινωνικές ε, συνθήκες προστασίας είναι πραγματικά φρικτές. Θα πρέπει να δούμε την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορείτε να βελτιώσει την κατάσταση πραγματικά. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θεωρώ ότι αποτελούν μια πλήρη λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αποτελεί φυσικά αυτό ένα σημείο εκκίνησης, ένα καλό σημείο εκκίνησης. Αλλά παρ' αυτά αυτές οι προτάσεις δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα των κοινωνικών προβλημάτων και τη ρίζα των προβλημάτων, του προβλήματος των συνθήκων εργασία. Θα θέλαμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι όλες αυτές οι προτάσεις ε, είναι αλληλοσυνδεόμενε. Και θα ήταν επικίνδυνο να αναλύσουμε και να επικεντρωθούμε σε μία από αυτές τις προτάσεις χωρίς να λάβουμε υπόψη και τις υπόλοιπε και τις συνέπειες που θα έχει στου υπόλοιπου τομεί. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις, οι εικονικές επιχειρήσεις δεν θα ε, απαλληφθούν πλήρως με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν έχουμε λοιπόν μια εταιρεία μέτρα στην, ε, στο Βέλγιο, με θηγατρική στη Ρουμανία, μόνο και μόνο για να μπορεί να απασχολεί οδηγού και έχει για παράδειγμα dispatching στην ε, Σλοβακία, η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά θα ε, καταφέρει να απαλείψει τη θηγατρική, αλλά όχι το κέντρο dispatching. Αυτό τι σημαίνει, ότι το κοινωνικό dumping και η έλλειψη ε, οδηγών και τα προβλήματα υγείας, έλλειψης κοινωνικής περίθαλψης, κοινωνικής προστασίας θα συνεχιστούν να υπάρχουν όπως και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρόνο ανάπαυση, η επιστροφή στην χωροκατοικία, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο. Χρειαζόμαστε ορισμό της κατοικία και μάλιστα ξεκάθαρα μέτρα για να ελέγχεται η επιστροφή, η πραγματική επιστροφή του οδηγού και επίση θέλουμε νομικέ διατάξει προκειμένου να υπάρχει αποζημίωση για την επιστροφή στην χώρα κατοικία από την εταιρεία. Δεν έχω χρόνο δυστυχώ να σα μιλήσω για τι προτάσει σε ό,τι αφορά τη μείωση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης 45 ώρων. Με την εξήγηση που θα μπορούσα να σας δώσω για την, να βοηθηθούν οι οδηγοί για να επιστρέψουν στον χώρο κατοικίας. Αυτή η ρύθμιση, επιτρέψτε μου να σας πω, Ό,τι και να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην οδογία για το, για το χρόνο εργασίας, το χρόνο εργασίας των οδηγών. Θα προσέξουμε λοιπόν ιδιαίτερα το στοιχείο αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απόσπαση. Είμαι απόλυτα, ε, αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτά που προτείνει για την απόσπαση των εργαζομένων. Είναι ευαίσθητο τομέα οι μεταφορές και έχουμε διάφορα είδη μεταφορών τα οποία αγγίζει η οδηγία αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν είναι κέρια σημασία οι, οι οδικέ μεταφορές να λάβουν την προσοχή που τους αρμόζει σε ό,τι αφορά την απόσπαση. Ποιε είναι λοιπόν οι προτάσει του ETF. Σε ό,τι αφορά τις εικονικές εταιρείε, ο μοναδικός πραγματικός τρόπος να τις καταπολεμήσουμε, ουσιαστικός τρόπος, είναι να υπάρχουν προδιαγραφές σε ό,τι αφορά το όχημα το οποίο θα πρέπει να οδηγεί και να κινείται, να κυκλοφορεί στη χώρα όπου έχει την έδρα τη εταιρεία. Ιδάλω δεν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε τι εικόνικε εταιρείε. Ό,τι αφορά το χρόνο ανάπαυση, θα πρέπει να είναι απαράλλαχτε οι ισχύουσε διατάξει. Και έτσι λοιπόν η εβδομαδιαία αναπαύση στα οχήματα θα πρέπει να απαγορεύεται και να φτάνει τα 45, 45 ώρες. Θα πρέπει να, συνεχίσουμε, να, να συνεχίσουν να ισχύουν οι εξαιρέσεις επίσης. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή τώρα στον χώρο α, κατοικίας, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα, γιατί θέλουμε να έχουμε μία, σα, ένα σαφή ορισμό του τι αποτελεί κατοικία. Γιατί είναι σαφές ότι αφορά τις δυνατότητες εφαρμογής ότι το κόστος, το κόστος ε, μετακίνησης θα πρέπει να καλύπτεται από την εταιρεία όπως και ισχύει και σήμερα σε ό,τι αφορά την απόσπαση. Θα πρέπει να υπαρχούν τομεακά μέτρα εφαρμογής και μάλιστα συγκεκριμένα για τις οδικές μεταφορές. Αλλά μέχρι εκεί μόνο μέτρα εφαρμογής τομεακά για τον τομέα των οδικών μεταφορών για μας δεν συζητάμε καν. Ναι. Να βγει ο τομέα των οδικών μεταφορών από την, ε, το πεδίο εφαρμογή τη είχε για την απόσπαση. Η απόσπαση μπορεί να ελέγχεται και μάλιστα αποτελεσματικά από τους εφείς Και ακούσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους ε, βουλευτές να μας λένε ότι είναι αδύνατο να φανταστούν ότι αυτή η τα ε, ταχογράφη θα είναι για όλα τα οχήματα μέχρι το 2034 και να υλοποιηθούμε έτσι. Αυτό χρησιμοποιήθηκε ως ε, λέξη. Εμείς ζητούμε αυτοί οι τα τα να, να εγκατασταθούν δύο χρόνια μετά την την ε, δημοσίευση του στην θέση του στην αγορά τον Ιούνιο του 2019. Μπορούν λοιπόν αυτοί οι ταχογράφοι να βοηθήσουν τον καλύτερο έλεγχο του Καμποτάζε. Υπάρχει και το ε, ηλεκτρονικό SMR, για παράδειγμα, CMR, το οποίο επίσης αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλουμε οπωσδήποτε, και θα κλείσω εδώ, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το οποίο διακήρυξε πριν από κάποια χρόνια ο πρόεδρος Γιούγκερ. Ίση αμοιβή για ίση εργασία στο ίδιο μέρος. Νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε μια εξαγγελία πάρα πολύ σημαντική και τώρα ο ETF περιμένουμε να το δούμε να Να συμβαίνει και είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεργαστούμε με κατανοητικό τρόπο προκειμένου η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και των υπηρεσιών να μπορεί να γίνεται με σωστό και ειρηνικό και ομαλό τρόπο σε όλη την Ευρώπη και να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι τα ίδια δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Παρίλο. Να ακολουθήσει ο κύριος Βρόνσκι, πρόεδρος Transport and Logistics της Πολωνίας. Έχει το λόγο κύριε. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την ε, Πολωνική Ομοσπονδία Ενώσεων Transport and Logistics. Είμαστε μια οργάνωση επιχειρήσεων και έχουμε πάνω από 25.000 εργαζομένους. Θα σας πω λίγα λόγια για τις ε, κοινωνικές συνθήκες της εργασίας καθώς και για τη δέσμη μέτρων κινητικότητας και την άποψή μας, αν πραγματικά λύνει τα προβλήματα ή όχι. Και πρώτο, ας εξετάσουμε πώς έχει εξελιχθεί η οδική μεταφορά από τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Ανά δεκαετία έχουμε ένα τεχνολογικό άλμα. Οι συνθήκες εργασίας βελτιώνονται διαρκώς και ίσως στο προσεχές μέλλον η εργασία των ίδιων των οδηγών ε, φορτηγών αυτοκινήτων να γίνει τηλεεργασία. Δηλαδή μπορεί να κατευθύνουν ίσω τα φορτηγά αυτοκίνητα από το σπίτι του. Οι συνθήκε εργασία, είπα και πριν, βελτιώνονται διαρκώ. Σα υπενθυμίζω ότι οι συνθήκε εργασία δημιουργούνται από τις μεγάλες επιχειρήσεις μεταφορών, οι οποίες προσπαθούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα που επιβάλλει ο νόμος. Ας εξετάσουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Εδώ θα συμφωνήσω βεβαίως με τον κύριο Παρίλο που μίλησε μόλις πριν λίγο. Πρώτον είναι ο κίνδυνος από την πλευρά της ασφάλειας. Υπάρχουν και βαριά ατυχήματα, υπάρχουν και επιθέσεις ε, κατά των φορτηγών αυτοκινήτων και των ε, οδηγών. Υπάρχει και το πρόβλημα των ελλείψεων ε, χώρων σταθμεύσεως. Λείπουν τουλάχιστον 30.000 χώροι στάθμευσης στην Ευρώπη. Ή υπάρχουν χώρε στάθμευσης οι οποίοι δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένοι με τουαλέτες κλπ. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν παρά μόνο μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό αποτελεί κίνδυνο και για τους οδηγούς αλλά και για το εμπόρευμα που μεταφέρουν στα φορτηγά αυτοκίνητα. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι και η μεταφορά εμπορευμάτων ανάμεσα στα δύο, σε δύο ε, περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάτι τέτοιο χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Ας δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Υπάρχει συχνά ε, δυσκολία στην κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους, δηλαδή υπάρχει πολύ πυκνή κυκλοφορία. Υπάρχει είναι, είναι, δυνατόν, είναι δυνατόν υπό τις συνθήκες αυτές να εξασφαλίζεται η ανάπαυση του εργαζόμενου μέσα στην καμπίνα του οχήματος. Ξαναλέω, ε, οι δυσκολίες κυκλοφορίας και αυτές οι εχμές είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από τη Βαρσοβία μέχρι τις Βρυξέλλες είναι 1350 χιλιόμετρα. Και σε κάθε περίπτωση που το κάνω αυτό, γιατί εγώ οδηγώ το αυτοκίνητο, περνάω τουλάχιστον ένα τρίωρο σε ε, σημεία κυκλοφοριακής αιχμής. Επομένως, οι κυκλοφοριακές αυτές αιχμές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, δεν υπάρχουν χώροι ε, για να αναπαυθεί κανείς, να κοιμηθούν οι οδηγοί. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Το, οι μέτρων κινητικότητας, το πακέτο κινητικότητας πιστεύω ότι θα ε, οδηγήσει και σε νέα προβλήματα. Είπαμε ήδη ότι οι καμπίνες των οδηγών για την ώρα είναι πολύ καλά εξοπλισμένες, των ε, φορτηγών αυτοκινήτων δηλαδή. Σε φτωχότερες χώρες, μάλιστα, τα φορτηγά αυτοκίνητα είναι μάλιστα καλύτερα εξοπλισμένα από ότι στα φορτηγά των ε, πιο εύπορων ε, δυτικών χωρών. Επομένως, οι ορισμοί που περιλαμβάνει το πακέτο κινητικότητας δεν το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Οι κουκέτες των οδηγών είναι καλύτερες από τους άλλους χώρους καταλήμματος και ανάπαυσης που προσφέρονται. Όλοι εδώ στην Ευρώπη μιλούν για την ισότητα. Βεβαίω χρειαζόμαστε ισότητα, χρειαζόμαστε ίση μεταχείριση, δηλαδή ίσο μισθό για ίδιο μισθό για την ίδια εργασία. Παντού. Αυτό είναι σαφέ. Σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει ο οδηγό να αμείβεται το ίδιο. Όμω, πώ θα λυθούν τα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη. Υποτίθεται ότι θα το πράξει αυτό η οδηγία περί απόσπαση εργαζομένων, που όμω αφορά μονάχα το 1% των εργαζόμενων. Πώς θα λυθεί λοιπόν το πρόβλημα όταν αφορά μονάχα το 1%. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μια δήλωση δημαγωγικού χαρακτήρα. διότι προσπάθεια εξίσωσης σε ένα σημείο οδηγεί σε έλλειψη ισότητας αλλού. Δύο οδηγεί, για παράδειγμα, πολωνικής επιχείρησης. Ο ένας κατευθύνεται στην Ισπανία και ο άλλος προς την Λευκορωσία ή την Ουγγαρία. Ο ένας οδηγός αμείβεται με 3.710 ευρώ. Ο άλλος οδηγός στην ίδια, με, κάνει την ίδια δουλειά, ε, ε κερδίζει μόνο 1.500 ευρώ. Μπορεί ε, ίσως να εξαλείψουμε αυτή τη διαφορά αμοιβή, αλλά θα προκαλέσουμε διαφορές αλλού. Τώρα, τα καθήκοντα των εργοδοτών, ποια είναι αυτά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πακέτου ε, κινητικότητας. Εμείς στο γραφείο μας εξετάσαμε τις γαλλικές διατάξεις, τις γαλλικές νομικές διατάξεις και τις ε, βάλαμε στο τραπέζι. Ασφαλώς ε, είναι μεγάλος ο όγκος των εγγράφων αυτών. Τώρα, μια μικρή επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση, πώς θα τα καταφέρει να ξεδιαλύνει αυτό το κουβάρι ε, νομοθετικών ρυθμίσεων. Εν τέλει, ποιες είναι οι επιπτώσεις Το εθνικό δίκαιο, οι εθνικές ε, νομικές διατάξεις είναι περίπλοκες. Το ίδιο είναι και το ευρωπαϊκό δίκαιο. δεν αποκλείεται κανείς από την εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Αυτό σημαίνει όμως επιβάρυνση των επιχειρήσεων που ε, δραστηριοποιούνται σε πλήθος αγορών. 80% των επιχειρήσεων μεταφορών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις ή μικροεπιχειρήσεις. Είναι πρώην οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων οι οποίοι πήραν ένα δάνειο από την τράπεζα για να ανεξαρτητοποιηθούν. Δηλαδή οι ίδιοι οδηγούν το φορτηγό τους αυτοκίνητο και καμιά φορά βοηθεί και η οικογένειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι οικογένειες, πώς θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις περίπλοκες αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν είναι σε θέση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι δυνατό να ε, προσαρμοστούν. Ας δούμε τώρα τη διαφορά των αμοιβών. Οι διαφορές αυτές δεν αποτελούν dumping. Κανένα δίκαιο δεν παραβιάζεται εδώ. Είναι ε, απλώς η φυσική συνέπεια των διαφορετικών ιστορικών ποριών των χωρών μας. Οι διαφορές αυτές ε, μειώνονται βεβαίω, διότι συγχρονιζόμαστε διαρκώ όλοι και διότι εργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά. Και άρα μειώνουμε τι διαφορέ μα. Και δεν θα πρέπει να επιβάλλονται όμω οι ρυθμίσει αυτέ αναγκαστικά. Και κάτι ακόμη. Ο τομέα των μεταφορών είναι τομέας κέρια σημασία για τις οικονομίες, όπου όμως λείπουν πολλοί οδηγοί. Στην Πολωνία μας λείπουν 4.000 οδηγοί. Κάθε οδηγός μας μπορεί να αλλάξει εργοδότη πολύ γρήγορα. Ο εργοδότης όμως για να προσλάβει άλλον οδηγό χρειάζεται ένα μήνα να ψάχνει. Άρα οι νέες διατάξεις, οι νέες ρυθμίσεις συνεπάγονται τον κίνδυνο να υπάρξει αταξία στο περιβάλλον. Το πακέτο, των, το πακέτο κινητικότητας μπορεί να πετάξει έξω από την αγορά αυτούς που υποτίθεται ότι επιθυμεί να προστατεύσει. Δεν πρόλαβα δυστυχώ να τα πω όλα όσα θα ήθελα, αλλά πάντως σα ευχαριστώ που με επιτρέψατε να εκφράσω την άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βρόνσκι. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Χαρτ από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Μεταφορών Εμπορευμάτων, Εφοδιαστικής και Αποκομιδής Απορριμμάτων ή Αποβλήτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Πρώτα λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση την οποία ευχαρίστως αποδεχτήκαμε θα προσπαθήσουμε ε, να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα από τη γερμανική σκοπιά. Πρώτα όμως κάτι σχετικά με την ένωσή μας. Ένωση Ομοσπονδιών που εκπροσωπούμε περίπου 7.000, 7.000 επιχειρήσεις με πολλές χιλιάδες οχήματα και οδηγούς. Είμαστε λοιπόν η Ένωση των Ομοσπονδιών των Ενώσεων, των ε, Σωματείων ε, Μεταφορών. Αντιμετωπίζουμε πολύ σωματικές προκλήσεις, όλη δηλαδή η αγορά των μεταφορών. Καθημερινά λαμβάνουμε πληροφορίες από τα μέλη μας που μας λένε ότι ο συγκεκριμένος τομέας έχει φτάσει στο όριο της δυναμικότητάς του, καταλήγουμε σε καθυστερήσεις των μεταφορών και μας ζητούν πληροφορίες όσο το δυνατόν νωρίτερα για τις ε, διάφορες παραγγελίες που ε, θα πρέπει να έρχονται. Όχι μόνο οι δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις θίγονται από τα προβλήματα. Ενώσεις επιχειρήσεων και εργοδοτών και από την Ανατολική Ευρώπη παραπονούνται για ελλείψεις οδηγών. Αν δεν κάνουμε τίποτα θα αντιμετωπίσουμε συνολικά στην Ευρώπη ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι δεν θα βρίσκουμε οδηγούς δεν θα βρίσκουμε επαγγελματίες οδηγού Και αν δεν έχουμε τους συνεργάτε αυτούς, ένα σημαντικό μέρος τη οικονομία μας θα αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα. Εν ώψη του ιστορικού αυτού, ζητούμε να υπάρξουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και επίσης πολύ σημαντικό ένα κοινωνικά δίκαιο περιβάλλον, εναρμόνιση των ε, προτύπων και των ρυθμίσεων για τους ε, μισθού και για τι κοινωνικέ εισφορέ κλπ. Ασφαλώς εδώ μπορεί να βοηθήσει ο ηλεκτρονικός ταχογράφος. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι θα πρέπει ταχύτατα και όσο πιο αποτελεσματικά είναι δυνατόν να εισαχθεί το εργαλείο αυτό κοινέ συνθήκες για την εργασία που θα προσελκύσουν ιδίω τους νέους ανθρώπους να ασκήσουν το επάγγελμα του επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου, φορτηγού δηλαδή. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη, για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά. Κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται 30.000 οδηγοί και εκπαιδεύονται μονάχα 15.000 επαγγελματίες οδηγοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μείωση κατά το ίμιση. Ταυτόχρονα διπλασιάζονται τα πακέτα που ζητάει ο κόσμος να πάνε σπίτι του. Αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το πρόβλημα. Τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε την εξέλιξη αυτή. Η ευρωπαϊκή απελευθέρωση από την δεκαετία του 90 και μετά οι νέες εντάξεις, η διεύρυνση δηλαδή με 12 νέες χώρες μέλη, τα δύο αυτά οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του καθημερινού όγκου των μεταφορών. Ιδίω οι διαφορέ μεταξύ ε, μισθών ανάμεσα στην στην Ανατολική Ευρώπη είναι τεράστια. Πρόσφατη γαλλική μελέτη καταδεικνύει σημαντικές διαφορές στους ακαθάριστους μισθού. Από 300 ευρώ μέχρι 3.300. Το ίδιο για τις κοινωνικέ φορές. Από 670 ευρώ στη Βουλγαρία μέχρι 16.000 στο Βέλγιο. Για έναν οδηγό, για όλους τους οδηγούς ε, το ίδιο. Το κόστος ανά είναι 16.000 για έναν Ρουμάνο οδηγό, 56.000 ε, για έναν Βέλγο οδηγό. Δεν συμφωνώ βέβαια με όλα όσα είπε ο προλαλής σας. Δεν είναι φυσική αυτή η διαφορά. Οι εργοδότες μετεγκαθιστούν μεγάλους τόλους φορτηγών αυτοκινήτων. Μέχρι τώρα όμως προφόρμα, δηλαδή βάζουν στα φορτηγά καινούριου αριθμούς αυτοκινήτων, όμως εξυπηρετούν τους ίδιους πελάτες και κυκλοφορούν στα ίδια δρομολόγια, με πινακίδες αλλοδαπής βεβαίω. Όλα αυτά συμβαίνουν με, κάνοντας εκμετάλλευση των διατάξεων της οδηγίας περί εργαζομένων. και μπορούν έτσι να λειτουργούν με πολύ ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Το αποτέλεσμα όμως είναι μια άνηση κατανομή του ανταγωνισμού και χαμηλότερες αμοιβέ, χαμηλότερες κοινωνικές εισφορές που τελικώς ξεσπούν στις πλάτες των εργαζομένων και που ενισχύει ακόμα περισσότερο την αποχώρηση των οδηγών. Ακραίο παράδειγμα, ίσως είναι γνωστό, μια λετονική επιχείρηση η οποία προσλαμβάνει Φιλιππινέζους οδηγούς και τους στέλνει να κυκλοφορούν και στην ε, Βόρεια Γερμανία και στη Δυτική Ευρώπη. Τι ακολουθεί από αυτήν την εξέλιξη της αγοράς, με συγχωρείτε μια στιγμή, άλλο παράδειγμα, επιχείρηση Ανατολικής Ευρώπης προσφέρει, τα, ε, δηλώνει μάλλον τα φορτηγά του από άλλη χώρα. 1.200 από τα φορτηγά αυτά λειτουργούν διαρκώς στην Γερμανία. Άλλες εκατοντάδες τέτοια φορτηγά στη Γαλλία. Δεν θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Χωρίς να είναι καταχωρισμένα τα φορτηγά αυτά εκεί όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους. Δεν ασκώ κριτική σε καμιά επιχείρηση συγκεκριμένα, αλλά αυτό είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθούν πολλές επιχειρήσεις. Σας ε, δείχνω εδώ μια τμήμα από μια εφημερίδα. Εκπροσώπηση συνδικάτων οδηγών στην ρουμανική Τιμισοάρα, η οποία άνοιξαν γραφείο εκεί για να υπάρχει ένα συνομιλητής για τους Ρουμάνους οδηγούς. Χάνουν λοιπόν μερίδια αγοράς οι δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις γιατί αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό, από την άλλη μεριά οδηγούνται οι οδηγοί σε όλο και δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας. Βεβαίως, στην πράξη βλέπουμε και άλλα πράγματα. Σποραδικά επανέρχονται στις αιστείες τους οι οδηγοί. Συχνά λείπουν εβδομάδες και μήνες. Επομένως εκεί διακυβεύονται οι ώρες ανάπαυσης είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται στους χώρους στάθμευσης στους αυτοκινητοδρόμους και εκεί συμφωνώ απόλυτα με τους προηγούμενους ομιλητές δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες εργασίας. Χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις. Αυτό το τονίζει και η είδηση που βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια με φωτογραφίες από βαριά οδικά ατυχήματα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία με ε, αποτέλεσμα θανάτους οδηγών τα πράγματα επιδεινώνονται ακόμα με την, περισσότερο με την κατάσταση στους χώρους στάθμευσης. Απάνθρωπες συνθήκες στους χώρους στάθμευσης που οδηγούν και σε σημαντικό κίνδυνο απόψη ασφάλειας. Ποιες είναι λοιπόν οι κεντρικές απαιτήσει της ε, Ένωσης μας. Χρειαζόμαστε έντιμο ανταγωνισμό, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς, τέλος στο κοινωνικό dumping, πραγματική εφαρμογή της ε, οδηγίας για απόσπαση εργαζομένων, ευφυής ταχογράφος, ηλεκτρονικός ταχογράφος, παραπέρα απελευθέρωση ιδίως στις διατάξεις του Καμποτάζ θα πρέπει να επιτραπεί μόνο εφόσον υπάρχει, υπάρχει εξίσωση των κοινωνικών διατάξεων, όχι πριν, ποτέ. Οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση στην αγορά και στο επάγγελμα θα πρέπει να ισχύουν για όλους όσους συμμετέχουν στην αγορά και για όλες τις κατηγορίες αχημάτων και για οχήματα κάτω των 3,5 τόνων συνολικού βάρους, τέλος της κατάχρησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών για την κατάχρηση σε βάρος των σχετικών διατάξεων, η κυκλοφορία στην Ευρώπη. η γύρι δηλαδή που κάνει το φορτηγό αυτοκίνητο θα πρέπει το αργότερο σε τρει ή τέσσερι εβδομάδε να οδηγούν να επιστρέφει στην βάση του. Δεν θα μπορούν να ε, παραμένουν φορτηγά αυτοκίνητα σε ε, δημόσιους ε, χώρους στάθμευσης. Χρειάζονται ηλεκτρονικές, ε, ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου και με σοβαρότατους ελέγχους, αυστηρότατους ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων. Διότι θεωρούμε ότι παρόλες τις σωστές εν μέρη νομοθετικές διατάξεις, η κατάχρηση οργιάζει διότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Engelhardt και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ροντρίγκε Μεντάλ που είναι διευθυντής της Confibas του Συνδέσμου Εταιριών Λεωφορείων. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το μου επιτρέπετε να σας μεταφέρω τις απόψεις ε, του τομέα των οδηγών λεωφορείων ε, και καλή επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέβρεση λύσεων σε αυτό το τομέα. Όπως σας είπα, αντιπροσωπεύω τον τομέα των ε, λεωφορείων και για να σας δείξω μια εικόνα του τι αντιπροσωπεύει αυτό για την Ισπανία, έχουμε 3.500 ε, εταιρείε στην Ισπανία με ένα στόλο 42.000 λεωφορείων και καλύπτουμε και τις συνδέσεις ανάμεσα σε πόλεις και ε, χωριά στην Ιταλία. Έχουμε ένα τζίρο τριών δις ετησίως με ε, φορολόγηση 1,5 δις και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το λεωφορείο στην Ισπανία ε, μεταφέρει πάνω από 1,5 ε, εκατομμύριο κόσμο ετησίως ε, είναι τεράστιος αριθμός και οι συνθήκες οι κοινωνικές και των, οδηγών μας και των εργαζομένων μας θεωρούμε πολύ, ε, πολύ σοβαρά υπόψη γιατί είναι και η εικόνα μας ο οδηγό είναι αυτός που έρχεται σε άμεση επαφή με το ταξιδιώτη όταν εκείνος μπαίνει στο λεωφορείο. Είναι ο εκπρόσωπο τη εταιρεία μα. Εγώ πέρυσι συμμετείχα σε μια μελέτη, μια μελέτη που έγινε από το Ίδρυμα Φρανσίσκο Φορέλ για τι οδικέ μεταφορέ στην Ισπανία και κάνει αναχώρα μια σύγκριση του νομικού συστήματο που διέπει του οδηγού και του οδηγού στα δημόσια μέσα μεταφορά ε, αναχώρα. Αναλύει επίσης ε, τα συνδικάτα, το δικαίωμα σε απεργία, αν πρέπει να το κάνουν μεμονωμένα ή αν πρέπει να γίνει μέσα από τα συνδικάτα, πώς γίνονται συλλογικές διαπραγματεύσεις, αν η συλλογική διαπραγμάτευση είναι δεσμευτική σε εθνικό επίπεδο ή αν γίνεται σε κλαδικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές διαφορές, ακόμα και σε μια, μέσα στην ίδια χώρα οι συλλογικές συμβάσεις δεν έχουν, διαφέρουν διαφέρουν μεταξύ τους, πούμε και μέσα στην Ισπανία, από ένα μέρος στο άλλο της Ισπανίας, αλλά και στη Γερμανία, πούμε, στα διάφορα κρατήδια, οι συμβάσει, οι συλλογικέ προέβλεπαν διαφορετικές αμοιβέ, ας πούμε. Ε, οι διαφορές υπάρχουν λοιπόν όπως είπα στους μισθούς, στο χρόνο ανάπαυσης, ε, ακόμα και αν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Υπάρχουν όμως ε, διαφορές και εφαρμόζονται διαφορετικά σε άλλες ε, χώρες ε, το τηρούν κατά γράμμα, σε άλλες όχι. Εξετάσαμε και τις συμβάσεις σε κάθε χώρα. Η τροποποίηση των όρων μιας σύμβασης, ας πούμε σε κάποιες χώρες βλέπαμε ότι το να στείλει κάποιον οδηγό από το ένα μέρος εργασίας στο άλλο δεν σήμαινε καμιά αλλαγή στην σύμβαση. Σε ορισμένες χώρες ας πούμε μπορούσε κανείς ε, ε, να προσλάβει με 15 μέρες δοκιμαστική περίοδο, σε άλλες χωρίς περίοδο δοκιμαστική, σε άλλες ε, με μεγαλύτερη περίοδο και ούτω καθεξής. Στις διεθνείς μας ε, υπηρεσίες, όταν δηλαδή πάμε από την Ισπανία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα, όπως είπαν και οι υπόλοιποι εδώ ε, ομιλητές. Σε άλλες χώρες χρειάζεται να γραφτούν στους ε, εθνικούς καταλόγους, σε άλλες όχι, σε άλλες όχι. Και αυτό είναι πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές φορές ε, είναι αυτό μεγάλος γραφειοκρατικός φόρτος. Πολλές φορές δεν ξέρουν καν ότι πρέπει να γίνουν. Σε κάποιες χώρες πρέπει να υπάρχει νομική εκπροσώπηση, σε άλλες όχι. Σε ορισμένες χώρες ζητούν το έντυπο α1 για να μπορεί να μετακινηθεί ο οδηγός, σε άλλες όχι και ανάλογα με τις συμβάσεις ε, τις συλλογικέ, ναι, πρέπει να εφαρμόσεις ε, το ελάχιστη αμοιβή το μήνυμο μισθό. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα λέω για να πω με δύο λόγια ότι δεν είναι εύκολο για μια εταιρεία να κάνει τους λογαριασμούς και να κάνει τους υπολογισμούς όλους αυτούς. Έχουμε όμως και ένα κανονισμό που σημαίνει που είναι η πρόσβαση των ε, εταιριών στο διεθνή, στις διεθνείς υπηρεσίες μεταφορών με ε, λεωφορείο. Εκεί ορίζονται όλα. Όταν ε, υπάρχει, ας πούμε, μετακίνηση από τη χώρα προέλευσης σε μια άλλη χώρα και αφήνει εκεί επιβάτες, αν μεταφέρει από μια τρίτη χώρα σε τρίτη χώρα, αλλά περνώντας από κάποιο κράτος και ούτω καθεξής και Επίσης είναι πολύ καλά ρυθμισμένο το πότε μπορεί να γίνει καμποτάζ. Ας πούμε, ε, ας πούμε αυτό που λέμε ταξίδι με κλειστή πόρτα, όπως το λέμε. Ας πούμε είναι Μάιος, ε, τελειώνουν τα σχολεία και πάνε συνήθως ε, τα παιδιά ένα ταξίδι Ας πούμε στη Ρώμη, στο Παρίσι, ας πούμε ότι φεύγει ένα πούλμαν από τη Σαραγώσα στην Ισπάνια και πάει στο Παρίσι ή στη Λισαβόνα. Σε καμία στιγμή δεν παίρνει άλλους επιβάτες. Είναι μια υπηρεσία, όπως είπαμε, με κλειστές πόρτες και οι νόμοι λένε το εξής, ε, ότι δηλαδή πάει και έρχεται, αλλά από την άλλη πλευρά επειδή δεν αφήνει και δεν παίρνει επιβάτες, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι διεθνής υπηρεσία. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια προσπάθεια μακροπρόθεσμη και προσπαθεί να βρει λύσεις, Βλέπουμε ποιε είναι οι κοινωνικέ πτυχέ και προσπάθειε τη της όμω υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Για παράδειγμα, η πρόσβαση και η άδεια άσκηση του επαγγέλματο του μεταφορέα είναι πολύ συγκεκριμένη και σχετίζεται με την πρόσβαση στην άδεια μεταφοράς αγαθών και ταξιδιωτών. Αυτό το μήνυμα που σας, εγώ έχω να σας πω είναι ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση μεταξύ των τομέων γιατί άλλο τα αγαθά, άλλο οι ταξιδιώτες, άλλο οι άνθρωποι. Κάνουμε μεν μεταφορές αλλά μεταφέρουμε διαφορετικά είδη ας το πούμε έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και για την απόσπαση των εργαζομένων. Ο τομέας των μεταφορών είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι κινητός, κινούμενος. Δεν έχει νόημα να βάλουμε μαζί την αναθεώρηση της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους με τις διεθνείς μεταφορές. Καλύτερα είναι να κάνουμε πιο ειδική νομοθεσία για τις διεθνείς μεταφορές. Εμείς στον, υπο... στον τομέα των επιβατικών, των, επιβατικών, των μεταφορών επιβατών είναι κάπως πολύ διαφορετικό και έγινε και άλλη μια μελέτη που λέει ότι όταν ας πούμε από τρεις μέρες ε, ε, είσαι εκτός του, χώρα χώρας πρέλευσή σου και αυτός ο οδηγός θεωρείται αποσπασμένος, νομίζουμε πως είναι πολύ λίγος χρόνος γιατί Τελικά αυτό θα ζημιώσει τις δραστηριότητες των ε, υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείε μεταφοράς επιβατών. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα. πρέπει να δούμε τους χρόνους ανάπαυσης. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος ανάπαυσης γιατί ένας άνθρωπος που οδηγεί λεωφορείο με επιβάτες πρέπει να είναι καλό, ξεκούραστος, δεν μπορεί να πιέζεται. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που, πρέπει, που σας δίνω εγώ, ότι πρέπει αυτό να το λάβετε υπόψη. Δεν είναι το ίδιο οι οδηγοί που μεταφέρουν επιβάτες και οι οδηγοί που μεταφέρουν φορτία. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυφθούν υπόψη οι διαφορές. Είναι καλή προσπάθεια να βελτιωθεί η νομοθεσία, όμως να υπάρξει συντονισμό περισσότερο ανάμεσα στα κράτη-μέλη, να υπάρξει διάδοση των πληροφοριών, γιατί τελικά επειδή είμαστε σε μια χώρα περιφερειακή όπω είναι η Ισπανία, προσπαθούμε να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες αλλά και στις γειτονικές χώρες για ότι κάθε φορά οι οδηγοί μας πρέπει να περάσουν από αυτές όλες τις χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το λόγο και που μιλήσατε όλοι. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση. Ο κανόνας του παιχνιδιού είναι απλός. Κάθε ομιλητής θα έχει δύο λεπτά και θα είμαι αδιάλακτη για το χρόνο γιατί είναι μετρημένος για να μπορέσουμε να έχουμε τις απαντήσεις σας στις διάφορες ερωτήσεις των βουλευτών. Να ξεκινήσουμε από τον εισηγητή μας για την απόσπαση των εργαζομένων σε αυτό το πακέτο για την κινητικότητα της Επιτροπής Μεταφορών. Έχει η κυρία Μέρζα Κίλωνεν έχει τον λόγο που είναι η εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε tarjottu. Äh, käytän aikani muutamiin kysymyksiin. Να επικεντρωθώ σε αυτά που σχολιάσατε. Ποια είναι λοιπόν η δική σας αξιολόγηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τα αίτια της έλλειψης ε, ε, ελέγχου της εφαρμογής της τρέχουσας νομοθεσίας. Δεν τιμωρούμε τις επιχειρήσεις εκείνες που προβαίνουν σε παραβιάσει των διδάξεων. Επίσης, ε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε ό,τι αφορά τις ε, κυρώσεις που επιβάλλονται για την ε, παραβίαση συλλογικών συμβάσεων. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει απαραίτητα παρανομία, αλλά τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις που δεν σέβονται τους νόμους, ε, τιμωρούνται ή κατά πόσον επιβάλλονται κυρώσεις. Αυτό προφανώς η έλλειψη τέτοιων κυρώσεων προκαλεί συγκριτικό μειονέκτημα σε όσους ακολουθούν το γράμμα του νόμου. Τέλος, ένα στοιχείο το οποίο ανέφεραν και οι ομιλητές μας. Οι οποίοι δεν είναι καν στο επίκεντρο των προβλημάτων των οποίων προσπαθούμε να επιλύσουμε. Άρα, βράχει πρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα. Πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα και το πρόβλημα των, ε, του χρόνου ανάπαυσης. Ποιες είναι οι ελεκτικές λύσεις και πώς μπορούμε λοιπόν να λύσουμε το θέμα αυτό του χώρου και του χρόνου ανάπαυσης. Ευχαριστώ, Λαϊκή, κυρία Τέλη. Να δώσω την, το λόγο στην κυρία Λαμπόγιοβα. Έχετε δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η συγχύτρια της Επιτροπής Απασχόλησης για την Απόσπαση των Εργαζομένων ε, των Οδηγών, αλλά και ε, της έκθεσης που θα ψηφίσει ε, σε λίγο στην Επιτροπή Απασχόλησης και σας καλώ μάλιστα να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου σε ό,τι αφορά το φάκελο της ε, μεταφορών. Σε ό,τι αφορά την επερχόμενη ψηφοφορία ζητούμε σε ένα μη σκέψη να υπάρχει στον τομέα των μεταφορών ιδιαίτερη νομοθεσία σε ό,τι αφορά το επερχόμενο πακέτο για την κινητικότητα, αλλά έχουμε και κινητικότητα Έχουμε επίση τροπολογίε που ζητούν την εξαίρεση του τομέα των, των μεταφορών. Και ζητούμε και ειδικέ διατάξει μέχρι ότου στο ενδιάμεσο διάστημα πριν από την εφαρμογή του πακέτου κινητικότητας. Ε. Και επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό, θα μπορούσα να μιλήσω ώρες. Αλλά δύο θέματα είναι πιο σημαντικά. Καταρχάς, η εφαρμογή. Μα όπω και σε όλου του κλάδους και στις μεταφορές, το προβλήματα ξεκινάνε από την ελληπή εφαρμογή. Γιατί πάντα θα υπάρχουν εταιρείε που ε, προβαίνουν σε ενέργειες που αποτελούν απάτη. Θα πρέπει να είναι απλοί οι κανόνες, να μπορούν να τις εφαρμόσουν αυτοί που θέλουν να τις εφαρμόσουν. Πώς μπορούμε να βρούμε λοιπόν ισορροπία μεταξύ εφαρμογής και των νέων κανόνων, σύμφωνα με τους ομιλητές. Ποια πιστεύετε είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην παρούσα φάση. Δεν φτάνουν οι κανόνες ή δεν φτάνουν οι έλεγχοι. Να κοιτάξουμε, μην να μην προβούμε τελικά σε μέτρα προστατευτισμού στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει αυτό το όραμα της ενιαίας αγοράς και πρόσφατα κάποιες από τις προτάσεις των Ευρωπαϊκής δεν δίνουν εντύπωση ότι ορθώνουμε πάλι σύνορα μεταξύ των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορεί λοιπόν ε, επίσης θα αποφύγουμε το υπερβολικό γραφειοκρατικό άχθος και για τους εργαζόμενους και για τις εταιρείες. Ευχαριστώ ο κύριος Βαντεκάμπ, ο οποίος είναι και ο εισηγητής ε, για το χώρο, το χρόνο ε, οδήγησης. δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει επιτρέψτε μου. Και για τους τέσσερι ομιλητέ. αλλά και κυρίως τον κύριο Έγγελχαρτ και την κυρία από το ETR. Ποιο θα πληρώσει το χώρο, το χώρο στάθμευσης. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Επιτροπή Απασχόληση ότι οι χώροι στάθμευση θα αποτελέσουν την νέα κοινωνική πρόκληση και τον κύριο από την Πολωνία να ρωτήσω, διατίθενται οι εταιρείε, προτίθενται να πληρώσουν και αυτέ ε, για του χώρου στάθμιση. Δεν φτάνουν οι επιδοτήσει. θα πρέπει να γίνουν και ιδιωτικέ επενδύσει. Αυτή η πρώτη ερώτηση λοιπόν. Ο ιδιωτικός κλάδος θα πληρώσει γι' αυτό. το δεύτερο θέμα, ψηφιοποίηση. Διάβασα το φυλάδιο των Πολωνών επιχειρηματιών για το πώς ο τομέας των μεταφορών καταστρέφεται. Και το θέμα λοιπόν είναι μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο πολλά από τις διεκπαιρεώσεις διαδικασίες μας ε, ηλεκτρονικά. Λιγότερη ρύθμιση και πιο πολύ ψηφιοποίηση θα έλεγα. Και και έχω και καιρό να πω και το εξή. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ε, οι απειλές ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν στέκουν όλα αυτά που μα είπαν οι ομιλητέ για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και αυτό το απευθύνω και ω ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν χρειάζεται να το απαντήσετε εδώ όλα να μα πείτε, ε, νομίζω ότι δυσκολεύουμε πάρα πολύ τις μικρομεσαίε επιχειρήσει να συνεχίσουν τι διεθνεί του μεταφορέ. Και θα ήθελα α, μια ερώτηση να... την ερώτηση να την απαντήσει και εκπρόσωπο του ETF. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βιμφάντεν Κάμπ και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάρ, εισηγητή τη χρηματοδότηση για το χρόνο οδήγηση. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εσά, αγαπητοί ομιλητέ, για τι εξηγήσει που μα δώσατε. Νομίζω ότι διάφορα θέματα ανακύπτουν διαρκώ σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τι αναξιοπρεπεί συνθήκες εργασία, την έλλειψη των οδηγών, ε, την έλλειψη υποδομών θέματα επίσης ασφάλειας στο, στους χώρους αναπαύσης. Εδώ και χρόνια λοιπόν συζητάμε τα ίδια προβλήματα. Και να σας πω ειλικρινά, δεν βλέπω με τις νέες προτάσεις να ε, βελτιώνεται δραστικά η κατάσταση. και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζητούν μεγαλύτερη σαφήνεια και αυτό τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την νομοθεσία να μην υπάρχουν παραθυράκια και να τα οποία τα καταχράζονται οι διάφοροι. Μία ερώτηση λοιπόν προς τους ε, εμπειρογνώμονες σε ό,τι αφορά το θέμα της μείωσης του χρόνου ανάπαυσης. Εγώ πιστεύω ότι τίθεται και θέμα ασφάλεια στους δρόμους. Όταν λέμε ότι οι συνθήκες εργασίας από τη μία αποτελούν στόχο και η ασφάλεια στους δρόμους, εδώ υπάρχει μια σαφή αιτιώδη συνέφεια. Συμφωνούν οι εμπειρογνώμονες και μια άλλη ερώτηση σε ό,τι αφορά αν θέλετε, το image του κύριου, αν θέλετε, του όλου κλάδου. Είναι τόσο περίπλοκη η διαμόρφωση αυτού του κλάδου και είναι τόσο δύσκολη η όροι που ισχύουν για τον τομέα αυτό που τελικά νομίζω ότι προκαλείται μια μόνιμη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συμφωνούν οι υπεργνώμονε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπάρ και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Νίλσεν. Να, εδώ. Από την Επιτροπή μας, από την Επιτροπή Μεταφορών, είναι ο εισηγητής για την πρόσβαση στην αγορά. Έχετε το λόγο κύριε Νίλσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντα το εξή. Σύμφωνο με αυτού που λένε ότι πρόκειται για ένα πακέτο. Ή όλα ή τίποτα. Όλα είναι διασυνδεδεμένα και αλλοσυνδεόμενα. Και να πω ότι δεν έχει σημασία τι κανόνε θα εφαρμόσουμε, θα περάσουν, αν δεν εξασφαλίσουμε την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι ταχογράφοι, λοιπόν, αποτελούν σημαντικά ζητήματα και σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τι εικονικέ επιχειρήσει, το επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί το πρόβλημα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζουν οι οικονομικέ επιχειρήσει ποιο είναι, ελάτε σε εμά και θα αποφύγετε και τα κοινωνικά, και τις κοινωνικές εισφορές και τους φόρους. Δεν είναι επαγγελματικό αυτό ο τρόπο αντιμετώπιση. Φτάνει τώρα η πρόταση τη Ευρωπαϊκή επιτροπή ή δεν φτάνει. Άλλη ερώτηση, επόμενη πολλοί που ασχολούνται με διεθνείς μεταφορές, πολλές εταιρείε, αλλά και εργαζόμενοι μας αναφέρουν ότι όταν είναι κανείς στον κλάδο αυτό ξέρει ότι όταν φεύγει από τη χώρα του όταν φεύγει από τη χώρα του ξέρει ότι για να γυρίσει θα κάνει λίγο καμποτάζ. Γιατί η δεν μπορεί να έχει αποζημίωση για την επιστροφή του. Δεν είναι τρόπο όμω αυτό. Ε, συμφωνούμε γι' αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία, αυτή η συνδυαζόμενη οδηγία ε, έπαιξε το ρόλο που ήταν να παίξει, αλλά πλέον δεν ε, λειτουργεί πλέον. Φαίνεται ότι αυτό πηγαίνει από την αγορά. Χρησιμοποιούνται σε τρόποι μεταφορά και χρησιμοποιούνται για έναν σκοπό σήμερα, για να αποφευχθούν οι κανόνε, να παρακαμφθούν οι κανόνε του καμποτάζ. Πώς λοιπόν θα θέλατε να δημορφωθεί αυτή η οδηγία κόμπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να οριστεί εκ νέου. Πώς θέλετε εσείς να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίλσε, ο κύριος Φοντανέ. Η κυρία Φοντανέ. Η συγγήτρια για την γνωμοτότηση της Επιτροπής Επασχόλησης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους μας ε, για τις ε, εισηγήσει που έκαναν σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα και με τόσες αντιφάσεις όπως είναι αυτό. Όλοι έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον να εγγυηθούμε τις ίδιες εργασιακές συνθήκες και δικαιώματα στους εργαζόμενους, όμως εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα επηρεάσει και τη βιωσιμότητα των εταιριών ε, αυτού του τομέα και ειδικά τις μικρομεσαίες στον τομέα των αποσπασμένων εργαζομένων. Δεν νομίζετε πως θα ήταν δυσανάλογη εφαρμογή στους εργαζόμενους που μόλις περνάνε κάποιες ε, μέρες εκτός της χώρας τους και ότι μπορεί να δημιουργηθεί έτσι ένα διοικητικό άχθος πολύ σημαντικό. Οι ειδικοί μίλησαν για τρεις μέρες σε μια περίοδο ε, ενός μήνα. Αυτό είναι πολύ λίγο και ε, ούτε γίνεται τίποτα σημαντικό για τις ε, περιφερειακές χώρες. Όμως, τι σημαίνει σε μια περίοδο ενός φυσικού μηνός σημαίνει. Θα ήταν λογικό να υπάρχουν, να είναι μάλλον διαδοχικές αυτές οι μέρες. Ε, να είναι διαδοχικές ημέρες αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες μέσα στο μήνα που οι ε, οδηγοί ε, να ασκούν το επάγγελμά τους. Έπειτα η δυνατότητα καμποτάζ από την πρώτη μέρη νομίζετε πως δεν θα αυξήσει αυτό το κόστος εξαγωγών των εταιριών και από την άλλη πλευρά η κατάργηση της εξαίρεσης για τα οχήματα βάρους κάτω των 3,5 ε, τόνων σημαίνει ένταξη και του 71 ε, ε, και η εξαίρεση αυτή δεν θα πρέπει να ζημιώσει την εσωτερική αγορά ή τον ελεύθερο ανταγωνισμό θεωρείτε πως είναι σωστό, σωστή εφαρμογή αυτού του κανονισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου το περιθώριο κέρδους τους θα μειωθεί πάρα πολύ και σε πολλές περιπτώσεις θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση των οδηγών. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, οι ερωτήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Ε, για το κατά πόσο πιστεύετε ότι θα πρέπει οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις εταιρείες ε, ε, είναι πολύ αυστηρές και πρέπει να επιβληθούν. Μετά έγινε λόγος για χωροστάθμευσης, αν δηλαδή ο ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως οικονομικός μοχλός. Μιλήσαμε για τα ψηφιακά, την ψηφιακή τεχνολογία. Θα έχετε κι εσείς γύρω στα δύο λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας, στις ερωτήσεις που σας αφορούν, να είστε σύντομοι. Ε, παρακαλώ να ξεκινήσουμε με την κυρία Βάντερ Πέλτ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει έλεγχος, αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει έλεγχος, ίσως όχι αρκετός έλεγχος, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για τους επιθεωρητές να ελέγξουν, γιατί συχνά δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στα άλλα κράτη-μέλη. Όταν σταματούν ένα φορτηγό στον δρόμο μπορούν να δουν ένα περιορισμένο αριθμό στοιχείων και δεν μπορούν να πάνε στη χώρα προέλευσης του φορτηγού. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει αρκετή συμμόρφωση, σε ορισμένε περιπτώσει ναι, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε γιατί. Γιατί καταρχάς, οι κανόνες δεν είναι ξεκάθαροι Υπάρχουν πολλά, πολλές ελλείψεις στους ορισμούς, αυτό είναι, αυτό είναι το ένα, ο ένας λόγος και έπειτα οι κανόνες ερμηνεύονται διαφορετικά από τα διάφορα κράτη-μέλη. Σε σχέση με το ερώτημα του κ. Βαντερκάμπ για τους χώρους στάθμευσης. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει αρκετός χώρος αλλά δεν υπάρχει και επιχειρηματικό μοντέλο για τους ανθρώπους που θέλουν να αναπτύξουν ένα είδος τέτοιων ε, χώρων στάθμευσης. Αν δείτε στους δρόμους, ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις χώρο ή περιβάλλον που να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να σταθμεύσουν όλα αυτά τα φορτηγά και να υπάρχει και χώρος ανάπαυσης για τους οδηγούς. Δηλαδή δεν είναι που δεν θέλουν οι εταιρείε να το κάνουν, αλλά δεν υπάρχει χώρος για την ψηφιοποίηση. Δεν μπορείτε να είστε ενάντια στην ψηφιοποίηση, αλλά πρέπει να είναι αυτό δυνατόν για όλους. Και εδώ επαναρχόμαστε στο πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου πολλές μικρές εταιρείες, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης οδηγεί είναι δηλαδή στο δρόμο καθημερινά, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και πρέπει να κάνει αυτήν την, όλα αυτά τα διαδικαστικά το Σαββατοκύριακο που είναι πολύ δύσκολο. Και Κάτι ακόμα για την εικόνα. Ξέρουμε ότι η εικόνα των μεταφορών δεν είναι καλή, αλλά η έλλειψη οδηγών είναι πολύ σημαντική και οφείλεται κυρίως σε δημογραφικά προβλήματα. Και αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε. Δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εφαρμογή και έλεγχο. Όταν υπάρχουν 2 με 3% υποχρεωτική έλεγχη, το 97% πιθανότητε υπάρχουν να μην ελεγχθεί. Και όταν ο εργοδότη μου λέει, Ναι, εμένα όταν μου βάζουν ε, πρόστιμο 2.400 ευρώ, αλλά εγώ είχα ήδη κερδίσει 100 χιλιάρικα, ε, όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ζήτημα. Υπάρχουν δυνατότητες βεβαίως. Φυσικά και υπάρχουν. Έχουμε μία πανεπιστημιακή μελέτη. Λοιπόν, έχουμε ε, 30 που έχουν ελεγχθεί και έχουν πληρώσει ε, πρόστιμο. Ε, αλλά υπάρχουν άλλοι 70 που έχουν ελεγχθεί. Ε, θα πρέπει όλα αυτά να ψηφιοποιηθούν. Ναι, γιατί με τον έχω e e γράφω, υπάρχει σε άλλου τομεί, για άλλα οχήματα, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειε θα σταματήσουν μόνο τα οχήματα που δεν είναι εντάξει και τους ε, οδηγούς που παρανομούν. Αντί λοιπόν να σταματήσουν 170, 170 ε, φορτηγά θα σταματήσουν μόνο τα 30 που έκαναν παράβαση. Θα πρέπει λοιπόν να τεθεί το θέμα της δυσαναλογίας. Είναι σημαντικό. Και τώρα, Λύσεις υπάρχουν όπως είπα. Για παράδειγμα, η εκατοπροτέρων δήλωση που περιλαμβάνεται στον 1457 να γίνει ένα κεντρικό σημείο στην Ευρώπη που γίνονται οι προκαταρτικές δηλώσεις, οι προηγούμενες δηλώσεις, ώστε να ελέγχονται καλά και να μειωθεί κατά 75% και αυτό είναι σε μια έκθεση της Κομισιόν οι υπηρεσίες ελέγχου. Τώρα, αν το μέσα αυτό είναι ελκυστικό. ε, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνθήκε εργασία. Και η πυραμίδα ηλικιακή εξηγείται και από αυτό. Είναι προφανές ότι έχουμε τα όργανα, τα μέσα, μάλλον τα εργαλεία για να ελέγξουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο. Και ναι, κλείνω και με τον ΕΦΗ, ταχογράφο, θα πρέπει να τον επιβάλλουμε, θα πρέπει να υπάρξουν και κάποια μεταβατικά μέτρα που θα καταργηθούν όταν σε όλα τα οχήματα θα έχει εγκατασταθεί ο ευφυής ταχογράφος. Ο κύριος Βρόνσκι. Szanowni Państwo, jestem z zawodu prawnikiem, ale należę do tych nielicznych prawników, którzy nie wierzą, że za pomocą... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, συγκαταλέγω μεταξύ εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει κανείς την πραγματικότητα μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις. Και με τον τρόπο αυτό απαντώ ήδη σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που έγιναν. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, θεωρώ ότι σήμερα για το λόγο αυτό δεν γίνονται σεβαστές οι ρυθμίσεις. Το ερώτημα είναι, είναι λογικές οι ρυθμίσεις αυτές, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ή όχι. Διότι ο κανονισμός 303 του 16 λέει ότι ο, εάν ο οδηγός έχει λησμονήσει ένα από τα έγγραφα. Αυτό θεωρείται σοβαρή παραβίαση και έχει βέβαια κάποια ε, επιρροή στις στατιστικές. Τώρα, τα ωράρια των οδηγών και αυτά επηρεάζουν τις στατιστικές. Μήπως πρέπει να ορίσουμε διαφορετικά το θέμα αυτό, μήπως πρέπει να βάλουμε ας πούμε προδιαγραφές, για παράδειγμα, για τον θαλαμίσκο του οδηγού και αν πληρούνται οι προδιαγραφές αυτές τότε επιτρέπεται να αναπαύεται εκεί. Εάν δεν ικανοποιούνται οι προδιαγραφές αυτές, τότε θα πρέπει να αναζητείτε άλλο κατάλημα. Άλλο ερώτημα. Εάν αποκλειστούν τα οχήματα κάτω των 3,5 ε, τόνων μικτού βάρους, το ερώτημα, άλλο ερώτημα τώρα. Ποιο ρόλο παίζει η έδρα της επιχείρησης για την ασφάλεια. Μήπω πρέπει να θέσει κανεί όμω την ερώτηση διαφορετική, διαφορετικά. Μήπω πρέπει να οριστούν τα ωραία των οδηγών για αυτά τα οχήματα, τα κάτω των 3,5 τόνων μεικτού βάρους και να μπει και σε αυτά ο ηλεκτρονικός ταχογράφος. μήπω είναι πιο σημαντικό αυτό από την έδρα της επιχείρησης. Το άλλο ερώτημα τώρα, Ποιο θα πληρώνει του χώρου στάθμευση. Και εμεί στην Πολωνία αγοράζουμε τώρα γερμανικούς χώρους στάθμευσης, τους πληρώνουμε δηλαδή, για τα λεωφορεία και τα φορτηγά μας αυτοκίνητα για να μπορούν να πάβονται εκεί οι οδηγοί μας. Ορίστε, ευχαριστώ. Ε, ε, εσείς τώρα, ο κ. Έγκελχαρτ, και εγώ ήμουν οδηγός με όχημα 40 τόνων, 18 χρόνια σε επιχείρηση με 7.040 ε, άτομα ε, φορτηγά αυτοκίνητα. Γνωρίζω λοιπόν και την άποψη των εργοδοτών και την άποψη των εργαζομένων. Οι έλεγχοι πρέπει να θεσμοθετηθούν έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται. Και βεβαίως πρέπει και οι φορτωτές να ε, υφίστανται ελέγχους οι οποίοι και, οι εργοδότες γιατί πάντοτε αναζητούσαν τους πιο φθηνούς ε, οδηγούς. Τώρα κύριε Βαντερκάμπ, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν σε αυτό που λέτε κάποιες δυνατότητες, γιατί δεν αποσυνδέουμε το μήκος της καμπίνας του οδηγού από το μήκος του συνολικού οχήματος, ώστε να έχει περισσότερο χώρο ο οδηγός. Διότι η καμπίνα του οδηγού είναι το σπιτικό του πρέπει να έχει ωστόσο τουλάχιστον και χώρο προσωπικής υγιεινής, όπως υπάρχει και στα τροχόσπιτα. Ένα μέτρο παραπάνω καμπίνα οδηγού θα λύσει πολλά προβλήματα. Κάποιος ρώτησε μήπως είναι προβολικά πολλές οι Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι συγκεκριμένες οι Και γι' αυτό δεν μπορούν να ελεγχθούν σοβαρά και έτσι κάνουμε φαύλο κύκλο. Τώρα, οι ώρες ανάπαυσης. 24 ώρες ανάπαυσης και επιστροφή στην οικογένεια. Αυτό που ζητούμε. Και αυτό μου λένε πάντοτε οι οδηγοί μου. Θέλουν να περνούν χρόνο με την οικογένειά τους. Πρόβλημα εικόνας. Ο οδηγός έχει τρία προβλήματα τώρα. Η αποζημίωση δεν είναι επαρκής. Από την άλλη μεριά, οι συνθήκες, τουαλέτες κλπ. δεν είναι όπως θα έπρεπε. Και η νεότερη γενιά θέλει τουλάχιστον μια γενιά, μετά από κάποιε ώρες εργασίας να επιστρέφει σπίτι της, να βρίσκεται την οικογένειά τη. Αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με πιο συγκεκριμένου κανόνες. Η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων προβλέπει τρει ημέρε. Βεβαίω είναι σχετικά πολύ. Δεν μπορεί όμω κανεί να το καταργήσει αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία ε, Ντελή. Κύριε ε, Μεντάλ, εσεί παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Ρωτήσατε αν το πρόβλημα είναι η εφαρμογή των κανόνων. Όχι, δεν είναι μόνο η εφαρμογή, είναι και η ερμηνεία. Συχνά δευτερεύουσες, δευτερογενείς μάλλον εθνικές νομοθεσίες ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να επιτρέπονται οι έλεγχοι αν υπάρχουν πολλοί, αν υπάρχουν λίγοι, σε κάποιους ε, δεν υπάρχει ε, ομοιογένεια. Σε, στα, σε άλλο μέρος, σε κάθε χώρα μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι ε, και περισσότερες χειρώσεις και αλλού λιγότερες. Έπειτα, ρωτήσατε αν οι ευρωπαϊκοί κανόνες επιβάλλουν νέα σύνορα. Εγώ πιστεύω πως οι δέσμοι της κινητικότητας ε, του Μαΐου βασίζεται σε αυτά που κάνουν κάποιες χώρες ε, ούτε ή άλλως. νομίζω πω ε, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή τη που δημιουργεί νέα σύνορα. Υπήρχαν ήδη αυτά τα σύνορα, ήδη ετοιμάζονταν. Ε, εμείς, ας πούμε, στο τομέα των λεωφορείων έχουμε πρόβλημα με έλλειψη οδηγούς, επαγγελματίε οδηγούς χρειάζεται ειδική άδεια οδήγησης. Δεν είναι μόνο το θέμα του μισθού, πρέπει να πληρώνται συγκεκριμένοι όροι, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που να καταστήσουν αυτό το επάγγελμα πιο ελκυστικό για τους νέους. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις ε, που εντάξει ήταν λίγο λακωνικές γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο αλλά η συζήτηση συνεχίζεται και θα δώσω αμέσω το λόγο. Θα κάνω μια ε, ανάμειξη ανάμεσα στους βουλευτές Επιτροπής Επασχόλησης και τους βουλευτές Επιτροπής ε, Μεταφορών και θα δώσω το λόγο στην κυρία Λουκασένσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι οι νομικές συντάξεις που προτείνονται προσαρμόστηκαν στις πολιτικές προσδοκίες. Δεν... Ε, ελήφθησαν υπόψη κάποιες πτυχές, όπως για παράδειγμα η πρόληψη των καταχρήσεων. Ακούσαμε ότι το διοικητικό αυτό θα αυξηθεί. Δηλαδή, αντί να δημιουργήσουμε θέσει εργασίας, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκαλεί μια κατάσταση όπου οι θέσει είναι όλο και πιο κοστοβόρε. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ποια θα είναι η επιρροή των νομικών διδάξεων τις οποίες εξετάζουμε στις θέσεις εργασίας. Έχω και μια ερώτηση να κάνω για τις εικόνικες αυτές εταιρείε. Γιατί να μην δημοσιεύσουμε ένα κατάλογο με τις εικονικές αυτές εταιρείε. Αν να δημοσίευση τη αμοιβή των οδηγών, γιατί να μην δημοσιεύουν και οι εικονικέ εταιρείε αυτά τα θέματα. Η κυρία Μόγα Σαρτιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ομιλητές μας έδειξαν πόσο πολύ αυτή η εργασία των οδικών μεταφορών είναι ιδιαίτερο τομέα. Θέλω να τους πω εγώ ότι στην οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους θελήσαμε να μην υπάρξει κενό, νομοθετικό κενό. Ε, τίποτα θα τα χειρότερο από το να αφήσουμε ένα τέτοιο ε, νομοθετικό κενό. Θα ήταν κάτι αντίθετο με τα συμφέροντα του τομέα και των εργαζομένων σε αυτόν και των εταιρεών. Εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα παραπάνω, αλλά νομίζω πως εδώ μπορούμε να πούμε πως αυτό το σημείο είναι θεμελιώδες σημασία. Κανένα στην Ευρώπη, καμιά εταιρεία και κανένας μισθωτός δεν θα έχει να κερδίσει αν αφήσουμε εδώ νομοθετικό κενό. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μωρέκ. Ξαρτιέ τώρα, Επιτροπή Μεταφορών, όπως είπαμε, όπως είπε και η Επίτροπος, η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους θα πρέπει να προστατέψει όλους τους τομείς και κυρίως το τομέα των μεταφορών. C'est Λοιπόν, συνεισηγητής Μιλήσατε για έλεγχο. Συμφωνώ μαζί σας για το θέμα του ταχογράφου. Βέβαια περιμένουμε το 2034, θα πρέπει να πάει πιο γρήγορα. Ναι, ένα διαδικαστικό έχω να κάνω, πρόεδρε, γιατί νομίζω πως είστε πρόεδρος και θα πρέπει να είστε ουδέτεροι. Παρακαλώ να απέχετε κριτικών παρατηρήσεων ε, και έκφρασης προσωπικών απόψεων όχι, θυμίζω την θέση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ήταν σαφής γιατί την ακούσαμε για το πακέτο για την κινητικότητα. Ναι, αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαστε το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε ε, Βίνου εγώ να τελειώσω με αυτό που ήθελα να πω και αν θέλετε στο τέλος της συνεδρίας θα το συζητήσουμε. Ας μην καθυστερούμε τώρα. Λοιπόν, μας μιλήσατε για τους ταχογράφους, είπατε πως το 2034 είναι πολύ αργά, όσο γίνεται πιο γρήγορα τόσο καλύτερα θα είναι. Αλλά είναι και θέμα ψηφιακό και το ψηφιακό σήμερα με, με την ψηφιακή τεχνολογία μπορούμε να προγραμματίσουμε ή να αποπρογραμματίσουμε με τρόπο που μπορεί να μην συμφωνούμε απόλυτα. Ε, άρα λοιπόν το πραγματικό μου ερώτημα είναι πώς μπορούμε να επιβάλλουμε πραγματικά τον έλεγχο. Ο ταχογράφος μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Είστε έτοιμοι σήμερα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει έναν Ευρωπαίο αστυνόμο, αστυφύλακα μια ε, ένα ευρωπαϊκό οργανισμό για τις οδικές μεταφορές. Αυτά. Δεν έχω χρόνο για τίποτα άλλο και περνάμε στον κύριο Μπάλας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ε, είμαι από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και θα ψηφίσουμε σε μια ώρα για το θέμα αυτό και έχουν υποβληθεί και τροπολογίες για τις οδικές μεταφορές. Ελπίζω να μην υπερψηφιστεί γιατί είμαστε σε ένα νομοθετικό κενό όσον αφορά τους εργαζόμενους στον οδικό τομέα και θα ήταν πολύ βλαβερό για ολόκληρο τον τομέα. Έτσι λένε και οι συνάδελφοι για το θέμα των ελέγχων. Όχι, δεν υπάρχει κενό και το έχουμε ψηφίσει εδώ στο Κοινοβούλιο και θυμήσατε και εσείς σωστά κύριε ότι εδώ είναι το Ευρωκοινοβούλιο την επιθυμία μας για τη δημιουργία ενός οργανισμού για την εποπτεία των οδικών μεταφορών. Υπερψηφίσαμε μόλις είναι αυτό δυνατόν να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί ταχογράφοι καθώς και ένα ηλεκτρονικό μητρό για να μπορέσουν εκεί να, να, καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία για τους μεταφορείς και τους οδηγούς. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλάς. Η κυρία Γκραπίνη, εσείς έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι ε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τις παρεμβάσεις των ε, εμπειρογνωμονών και διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Υπήρξαν, είπατε λοιπόν, για ελεύθερη αγορά, αλλά μιλάτε και για περιορισμούς. Να, η πρώτη αντίφαση. Έχουμε την εσωτερική αγορά. Είμαστε όλοι μέλη της, ε, της, ε, μέλη της εσωτερικής αγοράς. Και εφόσον θέλουμε να έχουμε ελεύθερη αγορά, πρέπει να λάβουμε υπόψη την επικουρικότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ορισμός του όρου κοινωνικό ντάμπικ. Άκουσα πολύ φρικτά πράγματα, ε, ότι δηλαδή για μια χώρα ένας συγκεκριμένος μισθός θεωρείται κοινωνικό ντάμπινγκ. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε αυτό το πράγμα. Τι είναι κοινωνικό ντάμπινγκ, τι είναι επικουρικότητα. Οι ορισμένοι μιλούν για συνθήκες, ας πούμε, ένας εργαζόμενος που εργάζεται για ένα, μια μικρομεσαία επιχείρηση, της οποίας τα φορτηγά διανύουν 3.000 χιλιόμετρα. Πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες, τους κανόνες ε, ε, και τις εργασιακές συμβάσεις ανάμεσα στις εταιρείε και τους οδηγούς. Εάν πιστεύουμε πως οι νόμοι της αγοράς λύνουν όλα τα προβλήματα, τι κάνουμε σήμερα για την έλλειψη των οδηγών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντερντέλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως κοιόδης για την για το ΕΛΚ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, ακούγοντας τους εμπειρογνώμονές μας, ε, διαπίστωσα και κατέστησαν και ήδη σαφές ότι η Κομισιόν ακολουθεί λάθος δρόμο μέσα σε αυτή την πρόταση. Ε, όταν θέλει να υποβάλει τους οδηγούς στους κανόνες περί αποσπασμένων εργαζομένων. Αποσπασμένων Και επίσης ε, φαίνεται να, ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες ε, λεπτομέρειες για τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακούσαμε ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία όσον αφορά τη θέση των μικρομεσαίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, έχετε λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων στις μικρομεσαίες και πόσες θέσεις απασχόλησης θα τεθούν σε κίνδυνο λόγω αυτής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Κυρία Γεζοβιέσκα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, ναι, εγώ είμαι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για αυτή, την, ακρο... για την ακρόση και για ε, τις ωραίες, ωραίες παρουσιάσεις από πλευράς των εμπειρογνωμόνων. Σε κάθε, για κάθε 100 ατυχήματα, τα 30 συνδέονται με την κατάχρηση των κανόνων. Σημαίνει αυτό ελλείψεις ε, του δικαίου, ε, λάθος ή διαφορετική ερμηνεία ε, των κανόνων από πλευρά των κρατών μελών. Θα ήθελα αυτό να είναι πολύ ξεκάθαρο ώστε εδώ, ειδικά στο Ευρωκοινοβούλιο, προσέχουμε ιδιαίτερα το θέμα της σαφήνειας και της βεβαιότητας της νομοθεσίας. Θα πρέπει κάτι ε, να είναι κάτι αυτό που ισχύει και για τις ε, νομοθεσίες των μεταφορών. Μήπως υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος όγκος νομοθεσία που είναι πολύ περίπλοκος στον τομέα των μεταφορών. Επίσης παρουσιάσατε ένα σχήμα όσον αφορά την ιδιαίτερο χαρακτήρα και το περίπλοκο χαρακτήρα των οδικών μεταφορών. Έχετε μετρήσει ποιο είναι οι επιπτώσει για το κόστο τη διεθνή μεταφορά και πόσο εμεί οι καταναλωτέ θα πληρώσουμε για την εισαγωγή αυτή τη νομοθεσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία παρατήρηση. Το να, μιλάμε για προστατευτισμό όταν ε, μιλάμε για την, τα δικαιώματα, για την νομοθεσία που προστατεύει τους εργαζόμενους, και νομίζω ότι είναι κάτι το παράλογο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους, ε, την οδηγία για την απόσπαση των εργαζόμενων, νομίζω ότι θίγεται θέμα και του στο το οποίο αποτελεί μία ε, βασική παρανόηση. δεύτερη ερώτηση είναι πραγματικά τόσο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να οργανώσουν την ε, διαδρομή των οδηγών προκειμένου να έχουν ένα σωστό χώρο και χρόνο ανάπαυση εκτό τη καμπίνα του, εκτό του φορτηγού και να επιστρέφουν μία φορά το την μήνα στο σπίτι του. Και εξηγήστε μου και γιατί δεν χρησιμοποιούνται τα επιτηρούμενα πάρκινγκ ή χώρε στάθμευσης και γιατί τελικά ξεχυλίζουν τα υπόλοιπα πάρκινγκ. Πώ γίνεται να υπάρχει χρηματοδότηση για τα επιτηρούμενου χώρου στάθμευσης και να μην χρησιμοποιούνται επειδή χρειάζεται να πληρώσουν αφού προσφέρουν όλου του όρου για να υπάρχει σωστή αναπαύση και τουαλέτες και ντους και ό,τι χρειάζονται και σε ό,τι αφορά την επιτήρηση των ε, φορτηγών. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά την περίοδο του καμποτάζ, ε, πιστεύετε ότι θα καταπολεμούσαν οι προτάσεις αυτές τα προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το καμποτάζ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πυρικόλα. Ευχαριστώ πρώτα και πρωτού θέσω τις μου να θέσω ένα γενικό σχόλιο που αποτελεί, θα έπρεπε να αποτελεί την ε, βάση της συζήτησης. Η ενιαία αγορά εξυπηρετεί τον κόσμο και όχι το αντίστροφο. Δεν εξυπηρετεί ο κόσμος την ε, ενιαία αγορά. Μιλάμε για βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί το σημείο κίνησης του Κοινοβουλίου και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά την υλοποίηση. Όλοι οι ομιλητέ μίλησαν για προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Άρα, μήπω χρειάζεται πιο πολύ συνεργασία μεταξύ των κρατών να υπάρχουν οργανώσει επίση επιθεωρήσεις εργασία ε, σε περιπτώσει που δεν τηρούνται οι κανόνε Για πείτε μα, τι πιστεύετε γι' αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ για ένα λεπτό. Ένα λεπτό λέω. Κυρία, ε, Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα θέλω να θέσω ότι μέσα σε αυτό το πακέτο υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας Ότι δηλαδή ο οδηγό του φορτηγού ή του λεωφορείου είναι ο υπεύθυνο για όλα. Δίνεται δηλαδή, αναθίθεται με υπερβολικά μεγάλη ευθύνη στον οδηγό, ενώ υπάρχει και ένας, ε, μια μαύρη λίστα για εταιρείε που χρησιμοποιούν κοινωνικό ντάμπινγκ, που έχει πολλές πολλές εκφάνσεις. Θα έπρεπε να κάνουμε ένα τέτοιο κατάλογο. κάποια οι περιφερειακές χώρες, γιατί ξέρουμε πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει πλάτος από την Πορτογαλία μέχρι την ε, Μαύρη Θάλασσα και από τη Φιλανδία μέχρι την απόλη και τη Φινισικελία. Αυτοί λοιπόν που είμαστε στην περιφερεια έχουμε προστεθέμενο κόστος ανά χιλιόμετρο που δεν το αφαιρούν αυτοί που είναι στο κέντρο. Κυρία Γιάλα Σάντερ, τελείωσε το λεπτό σα, λέει η πρόεδρο, Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Πώ λαμβάνετε υπόψη τι περιφερειακέ χώρε, και απίτα. Κυρία Γιάλα Σάντερ, δεν έχετε άλλο χρόνο, διακόπτη Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίτσελ Λούγκριν. Σας παρακαλώ να τηρείτε το χρονικό όριο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαντγκριν. Όπως ξέρετε, ήμουν 30 χρόνια οδηγός φορτηγού πριν μπω στο κοινοβούλιο. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα στη φορά τα σύνορα και πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές κοιμόμαστε καλύτερα στο φορτηγό από ότι στο ξενοδοχείο και όταν πρέπει να προστατεύσουμε και το φορτίο δεν υπάρχει πρόβλημα να δεν εκτερεύει κανείς ε, στο φορτηγό, αλλά το πρέπει να μπορεί κανείς ως οδηγός να μπορεί να επαναφάει, να μπορεί να κάνει να ντους όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος μέχρι να επιστρέψει στην οικογένειά του. Και αυτή η κατάσταση, ό,τι αφορά το καμποτάζ, δεν μπορεί να ελεγχθεί πλέον επαρκώς. Και βλέπουμε ότι πώς θα μπουν οι νέοι σε ένα κλάδο ο οποίος δεν λειτουργεί. Όλα είναι στραβά και ανάποδα. Πολλοί κόσμος επιστρέφει ε, και με και να φόρτηγα. Γιατί το καμπουτά τα έχει αλλάξει όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Είναι ο επόμενο μιλητή. Η πραγματικότητα είναι ότι οι κανόνε έτσι όπω έχουν δεν λειτουργούν. Έχουμε δανέζικε εταιρείε που ανοίγουν θηγατρικέ σε κράτη-μέλη με χαμηλού μισθού, μόνο και μόνο να μπορούν να κάνουν διεθνεί τέτοιε μεταφορέ. Αυτό που δεν ήταν ο σκοπό τη ενιαία αγορά, σε καμία περίπτωση. Πώ μπορούμε να επιλύσουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό του αθέμητου ανταγωνισμού, αν δεν υπάρχουν κανόνες σε ό,τι αφορά την απόσπαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ερτούκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και να πω και να ομολογήσω ότι κάπως έχω απογοητευτεί κι εγώ, γιατί εδώ και χρόνια οι εμπειρογνώμονες μας λένε τα ίδια και τα ίδια. Τις θέσεις τους επαναλαμβάνουν. Εγώ θα ήθελα πολύ παραπάνω οι εμπειρογνώμονες να μας κάνουν κάποια πρόταση κάποια στιγμή για το πώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον εκπρόσωπο της TIR. Είπατε ε, ότι θέλουμε ίσο μισθό για την ίδια εργασία. Όντω αυτή είναι η τοποθέτησή σα, γιατί υπάρχουν πολλοί από τι χώρε τη Κεντρική Ευρώπη και τη Ανατολική Ευρώπη που δεν προσυπογράφουν την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κίστελορ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Άκουσα με συμπάθεια. Αυτά. Ο κύριος Τέιλερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και άκουσα με συμπάθεια αυτά που ακούσαμε σε ό,τι αφορά τους τα ταχογράφους. Να πω το εξή. Μήπως ε, κάτι χάνουμε σε ό,τι αφορά την, την διαρκή παρακολούθηση των οδηγών. Έχουμε ένα τέτοιο μέσο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργοδότες ανά πάσα στιγμή και για τους μισθούς και την ανάπαυση και οι, οι αρχές εφαρμογές για να μην υπάρχουν περιπτώσεις απάτης. Γιατί λοιπόν χρειάζονται 15 ολόκληρα χρόνια για να εισαχθεί αυτός ο εφής ταχογράφος. Γιατί δεν μπορούμε να το εισαγάγουμε πιο γρήγορα και αν οι εταιρείε γλίτωνα και πολύ μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος με τους ταχογράφους αυτούς, δεν θα ήταν έξυπνο και και από οικονομικής άποψης. Ευχαριστώ και θα δώσουμε πάλι το λόγο, λέει η Πρόεδρος, για 20 δεύτερα στον κύριο Ερτούκ, ο οποίος δεν είχε καταλάβει πόσο χρόνο είχε στη διάθεσή του. 20 δεύτερα μόνο, κύριε Ερτούκ. Σας ευχαριστώ και ήταν όντω λάθος ε, διαχείριση του χρόνου. Έκανα την ερώτηση στον εκπρόσωπο του ELP Προ τον κύριο Παρίγιο να κάνω μια ερώτηση από το ETF τώρα. Όντω είναι πιο σημαντικό ο χρόνο ανάπαυση να είναι σε ξενοδοχείο, σε ένα στενόχρονο ξενοδοχείο ή ενδεχομένω σε σχέση με μια άνετη, αν θέλετε, καμπίνα του φορτηγού του κάθε οδηγού. Είναι πραγματικά αμετακίνητη η άποψή σα γι' αυτό. Ότι είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω, κύριος Ρικέ. Άκουσα τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων. Να διευκρινίσω το εξή σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, μάλλον το χάσμα μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης. Αμβλύνεται ή οξύνεται. Δεύτερη ερώτηση. βλέπετε ή οξύνεται. Δεύτερη ερώτηση. Οι εμπειρογνώμονε πιστεύουν ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού έχει να κάνει μόνο με το με τους όρους της εργασίας ή μήπως δεν πληρώνουμε επαρκώς τους οδηγούς αυτούς για την υπηρεσία που τους ζητούμε. Μόνο 30 δεύτερα κύριε Λεκέ, πάρα πολύ αποτελεσματικός ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Η μείωση του γραφείου κριτικού άχθους ε, μέσω της ε, νομοθεσίας. Αυτή είναι η συζήτηση και ο σκοπός της σημερινής συζήτησης μάλλον. Και συμφωνώ, συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γκραπίνη. Θέλετε να οριστεί το κοινωνικό dumping. Ίση εργασία για ίση δουλειά στον ίδιο χώρο απασχόλησης. Αλλά να το δευρύνουμε και να πούμε για παράδειγμα από τον ίδιο εργοδότη. Και τι θα σημαίνει αυτό στη συνέπεια. Μία άλλη ερώτηση προς τον κύριο Βρόντσκι. Είπατε ότι η απόσπαση εξαιρείται και ότι τρεις ημέρες δεν αρκούν. Πόσες μέρες λοιπόν αρκούν. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Zlotowski. Madame Demonté pour une minute. Σας ευχαριστώ πολύ. Από δική μου πλευρά, χώροι ε, στάθμευση. Να ρωτήσω του εμπειρογνώμενου αν είναι εφικτό και πρακτικό να υπάρξει μια παρέμβαση ε, με επιπληρωμή, ας πούμε μέσω project financing, με μια επένδυση από πλευρά ιδιωτών που μετά θα έχουν και κάποια έσοδα μέσα από τα ένισοδα που θα πληρώνουν οι, οι μεταφορείς. Έπειτα, Πώς θα λύσουμε τις διασυνοριακές μεταφορές. Εγώ έχω θέσει πολλές φορές αυτό το ερώτημα και δεν έχω πάρει απάντηση σε άλλες ευκαιρίες ακρόαση στην Επιτροπή Μεταφορών και πιστεύω πως το καμποτάζ μπορεί εύκολα να ε, ξεφύγει εάν υπάρχει ε, διασυνοριακή μεταφορά. Πώς μπορούμε λοιπόν από άποψη ρύθμισης να λύσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μίτεμπεργκ, ένα λεπτό. Έχω μια απλή ερώτηση, γιατί ακούμε ένα σωρό διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικές δηλώσεις. Η δική μου ερώτηση όμως προς τον Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οδηγικών Μεταφορών αλλά και ε, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων, την, τον τομέα μεταφορών, έχετε κοινωνικό διάλογο μεταξύ σας και μπορείτε να μας δώσετε ένα συμβαστικό κείμενο σε σχέση με αυτή την πρόταση, ώστε να έχουμε την απαραίτητο input από πλευράς και των δύο οργανώσεων, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τα απαραίτητα βήματα πριν να τελειώσει η εντολή μας, ώστε να βρούμε συμβιβαστικό κείμενο. Και έχω και μια έκκληση να κάνω προς τους συναδέλφους, γιατί ακούω πολλές δηλώσεις και λιγότερο ερωτήσεις, ενώ εδώ έχουμε ακρόαση. Χρησιμοποιείτε το χρόνο που έχουμε λοιπόν παρακαλώ στην Επιτροπή μας για να κάνετε τις δηλώσεις σας τις πολιτικές, αλλά στην ακρόαση ε, κάντε αυτό που πρέπει, δηλαδή να ακούσετε ε, και να θέσετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Βαρμίτεμπεργκ και τώρα στρέφομαι προς τους εμπειρογνώμονες. Έχετε δύο λεπτά έκαστος. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι πολύ, αλλά θα μπορούσατε ίσως να μας στείλετε και γραπτές απαντήσεις και μάλιστα έχουμε και διαφορετικές ερωτήσεις. Είστε όλοι υπέρ των ίσων ε, μισθών για ίση εργασία, για τα θέματα της, ε, του καμποτάζ. Ε, είστε υπέρ της ξεκούρασης της ανάπαυσης των οδηγών σε ξενοδοχείο ή σε καλά εξοπλισμένες καμπίνες. Χώρες ανατολικές και χώρες δυτικές. Τι γίνεται, λέει ο κύριος Ρικέ. Και ένα σωρό ωραίες και ξεκινώ από εσά, κυρία Βάντε Μπέλτ μου, για, ένα, για δύο λεπτά. Για τις επιχειρήσεις, τις εικονικές επιχειρήσεις, που είναι απλώς ένα γραμματοκιβώτιο, θα πρέπει να εξεταστεί ε, ε, συγκεκριμένα πρόκειται για κοινωνικό ντάμπινγκ και επειδή δεν υπάρχει και πραγματικός ορισμός του τι σημαίνει κοινωνικό ντάμπινγκ. Όποιον να ρωτήσει θα σας δώσει κάπως διαφορετικό ε, ορισμό για το τι σημαίνει κοινωνικό dumping, άρα θα είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανείς έναν ορισμό που να, εξυπηρετεί, ε, που να καλύπτει όλες τις απόψεις. Σε ό,τι αφορά τους χώρους σταθμεύσεως, πρόκειται για επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο δεν υπάρχει ακόμη. Υπάρχει έλλειψη χώρων και δεν είναι και πολύ, πολύ ρεαλιστικό βραχυπρόθεσμα να καλυφθούν δηλαδή όλα αυτά. Για τι ελλείψει οδηγών ρώτησε κάποιο γιατί υπάρχει ελλείψη οδηγών. Νομίζω ότι υπάρχει ένα απλό λόγο, βέβαια υπάρχουν και άλλε εξήγησει, αλλά πάντως μία απλή εξήγηση είναι το δημογραφικό. Υπάρχουν λιγότεροι νέοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι ή επιθυμούν να κάνουν τη δουλειά αυτή. Τέλο, όταν μιλούμε για κοινωνικό διάλογο, η UETR ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να συμμετάσχει στον κοινωνικό διάλογο και ευχαρίστως θα θέλαμε να βρούμε, να συμβαστούμε με τους συναδελφούς μας των συνδικάτων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό που να εξυπηρετεί όλους, αλλά και εμείς αντιμετωπίζουμε δυσκολίες μεταξύ επιχειρήσεων του Βορρά, του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης και όταν μιλούμε για ίση αμοιβή, για ίση εργασία, δεν ε, μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μπροστά στην βασική αιτία του προβλήματος που είναι η διαφορά στο εργατικό κόστος. Ακόμη και όταν ένας, εργα... ένας εργαζόμενος, ένας οδηγός δηλαδή, λαμβάνει την ίδια αμοιβή, το κόστος του για την επιχείρηση είναι διαφορετικό. Λόγω, ε, δηλαδή, εξαρτάται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ντέλη. Κύριε Παρίλο, εσείς παρακαλώ για δύο λεπτά. Εμείς ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού είμαστε υπέρ και έχουμε γράψει στην ΙΟΤΕΦ εδώ και καιρό και έχουμε καθορίσει και ορισμένα κριτήρια βασικού χαρακτήρα. Αρκετά σημαντικός φάκελος. Δεύτερο, οι αντιφάσεις ό,τι αφορά τον σεβασμό του δικαίου. Εμείς θέλουμε να γίνει σεβαστό το δίκαιο και η νομοθεσία. Τι λέει ο κανονισμός ΡΟΜ το εργατικό δίκαιο που εφαρμόζεται κατά περιφέρεια σημαίνει τον τόπο από τον οποίο ξεκινούν κανονικά οι δραστηριότητές μας. Και βεβαίως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λέει εφαρμογή του δικαίου, τίποτα άλλο. Τρίτο, ο συντονισμός για το καμποτάζ. Το μεγαλύτερο εργοδοτικό συνδικάτο των Ιταλών, Ανιτά, ε, ε, έγραψε έγγραφο ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτε περισσότερο από την άποψη της ψηφιοποίησης κλπ. Τώρα, για την ανάπαυση, χρόνος ανάπαυσης μέσα στην καμπίνα. Όχι, εβδομαδιαία ανάπαυση στο, στην καμπίνα, όχι. Η απόσταση, η μισθολογική απόσταση μεταξύ Ανατολής και, και Δύσης μεγαλώνει. Πρόκειται για μελέτη της CES δεν πληρώνουν αρκετά, γι' αυτό και δεν υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίε οδηγοί φορτηγών, είναι ένα από του σημαντικού λόγου. Και μπορώ επίση και να πω όταν του πληρώνουν, γιατί καμιά φορά η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική. Κοινωνικό διάλογο, κάνουμε προσπάθεια, έχουμε και μεγάλη συνάντηση που βλέπετε στι 27 Οκτωβρίου και θα προσπαθήσουμε οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι να τροφοδοτήσουν το διάλογο. Εμεί ω ΕΤΕΦ το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο να συνεχίσει να γίνεται είναι να εξετάσουμε και τις διασυνοριακές μεταφορές, που ήταν μια από τις τελευταίες ερωτήσεις σας. Βεβαίως η δυσκολία ξεκινά από τους ελέγχους και από τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων κρατών και των διαφόρων φορέων ελέγχου, που δεν υπάρχει ακόμα συντονισμό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς κύριε Βρόνσκι, δύο λεπτά πώς πάντα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή ε, Πρόεδρε για τις επιχειρήσεις γραμματοκιβωτίου. Γιατί να μην δημοσιεύω τα ονόματά τους, εμείς είμαστε υπέρ. Μπορεί να είναι 1500, μπορεί να είναι 300. Και τι κάνουμε, για χάρη τους αλλάζουμε ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο. Το αποτέλεσμα είναι σοβαρές ε, επιπτώσεις στην αγορά. ο ανταγωνισμός για τη μεταφορά εμπορευμάτων και η περιφέρεια ή η χώρα στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση καθορίζουν την τιμή. Άρα θα μπορούσε έτσι να μειωθεί το κόστος. Τώρα, ε, οι σταχογράφη. E Εγώ έχω εργαστεί και στην πολωνική διοίκηση και είχαμε κάνει προσπάθεια τότε να τους εφαρμόσουμε θεωρητικά μπορεί να αποτελέσει απάντηση σε πολλά προβλήματα. Όμως, φάνηκε πολύ γρήγορα, πολύ καθαρά, ότι ε, πολλοί οδηγοί είναι ιδιαίτερα επινοητικοί, κάνουν hacking στους ε, ηλεκτρονικούς ταχογράφους, οι οποίοι δεν λειτουργούν μετά σωστά. Και για τον εκ των υστέρων εξοπλισμό, retrofitting δηλαδή, το ίδιο θα είναι το πρόβλημα. Τέλος, η πάυση της απόσπασης. Αυτό θα είναι το... η Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο υπολογισμού για τις 15 μέρες, αν δεν θεωρούμε ότι ένα λεπτό σημαίνει μια ημέρα, τότε μπορούμε να κάνουμε την εισαγωγή και μετά από 10 μέρες. Εμείς ε, διεξάγουμε διάλογο με τα συνδικάτα, με την Solidarnosc, με τους οδηγούς, που ε, συμμετέχουν στο Συνδικάτο Σολιδάρνος. Έχουμε μάλιστα προωθήσει ορισμένες πρωτοβουλίες, έχουμε προσκαλέσει και την ETF ορισμένες φορές, υπήρχαν όμως ε, συγκρούσεις, ε, έτσι μας είπαν δηλαδή, υποχρεώσεων. Και που σημαίνει δηλαδή ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας. Αυτό έτσι το ερμηνεύουμε εμείς. Για την ποιότητα τώρα της παροχής υπηρεσιών, εμείς προσφέρουμε τις ίδιες υπηρεσίες όπως και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Ε, εσείς κύριε Έγγελ Χάρτ, δημοσίευση των ε, εικονικών επιχειρήσεων μάλιστα. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων επίσης υπέρ. Διαφορά 40.000 ευρώ στις, στα μισθολογικά, τα είπαμε αυτά. Γιατί δεν τα καταφέρουν Κάποιος διακόπτει. Πολύ ευχαρίστω να τα πω αργότερα. Σε δύο λεπτά όμω είναι δύσκολο να απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα. 45 ώρε έλεγα γιατί δεν καταφέρνω να του στείλω σπίτι. Γιατί αυτό είναι ο πυρήνα του επιχειρηματικού του μοντέλου. Έξι μήνε έξω στην Αλουδαπή ο οδηγό για να είναι όσο γίνεται πιο φτηνέ οι μεταφορέ. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν και φυλασσόμενοι χώροι στάθμευση, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται παρόλο που υπάρχουν, γιατί δεν τα προβλέπει το επιχειρηματικό μοντέλο αφού πρέπει να πληρώσει για αυτού του χώρου στάθμευση. Αυτό που λέει ο Λούντγκρεν είναι σωστό και εγώ θεωρώ ότι εκτό από το μισθό πρέπει να παίξουν ένα ρόλο και οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες να επιτρέπουν τον σχεδιασμό της ζωής του καθενός. Κύριε Έρτουκ, Έχουμε κάνει ένα κεντρικό σχεδιασμό, ευχαρίστως να σας τον υποβάλουμε. Και έχουμε δώσει και απάντηση και σε κάθε ένα από τα, λεπτομερή, από τα λεπτομερή προβλήματα. Διάλογος, ανατολής δύσης. Βεβαίως και υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα, όμως διάλογος διεξάγεται και αυτό ε, μα οδηγεί να διαπιστώσουμε ότι και στην Ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουν πλέον επιχειρήσει τα ίδια προβλήματα που είχαμε εμεί 5-6 χρόνια. Έλλειψη οδηγών, τα είπαμε, ε, μισθολογικά και τη προσωπική ζωή. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Συνεργασία με την ETF. Εμεί συνεργαζόμαστε με την εθνική εκπροσώπηση, το Συνδικάτο Βέρντι στη Γερμανία. Συνεργαζόμαστε και με το ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα προτινόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ροντρίγκης μετά αλλά έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα για τα ερωτήματα που αφορούσαν τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό για να λυθεί το, λυθεί το θέμα των οδικών μεταφερών. Ναι. εγώ είμαι ε, οπαδός της ήπιας νομοθεσίας. Υπάρχουν πολλά μέσα για νομοθεσία, αλλά το πρόβλημα είναι ε, οι ε, διαδικασίες όταν υπάρχει παράβαση. Υπάρχουν διάφορες νομικές πράξεις ε, και διατάξει, Εμείς στα κρατημέλη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά ε, όλα αυτά για να μπορέσουμε να πούμε πώς ερμηνεύεται το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο. Τώρα, για το θέμα των Ε, περιφερειακών χωρών πολύ συχνά παραμελείται αυτός όταν ε, ρυθμίζονται οι διάφορες υπηρεσίες. Ίσως ας πούμε το ευρωπαϊκό, ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περισσότερο ότι δεν είναι όλες οι χώρες στην ίδια κατάσταση όταν θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή όταν κάνουν εμπορικές προσφορές. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο για δύο λεπτά για να ε, συνάξει τα συμπεράσματα και μετά θα κλείσω και εγώ, θα συνοψίσω και εγώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ε, ήταν μια συζήτηση για την αξιοπρέπεια, για τη συνεργασία, για τον ανταγωνισμό με χαμηλότερες φιλοδοξίες ή τον ανταγωνισμό ε, μέσω της αριστείας, γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο ανάμεσα σε κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταγωνιζόμαστε και με τον υπόλοιπο κόσμο. Και μπορούμε να έχουμε βιώσιμο ανταγωνισμό όταν ο κόσμος πιστεύει και γνωρίζει πως αντιμετωπίζεται με δίκαιο τρόπο και ότι δεν πέφτει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ε, άρα λοιπόν σε σχέση με όλα αυτά ήταν πολύ καρποφόρα ε, και ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ. Σύντομα θα κάνουμε και ψηφοφορία. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να λάβουμε υπόψη τα όσα ακούσαμε. Σας ευχαριστώ όλους που μας δώσατε την εμπειρία σας και τις σκέψεις σας για αυτό το πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια είναι είδη συμπεράσματος στο όνομα της Επιτροπής Μεταφορών. Εγώ θα κλείσω. Εάν εμποδίζετε θα ε, βγείτε από την αίθουσα. Είμαστε στην πρώτη σειρά κροάσεων. Είναι πραγματικά μεγάλη συμβολή στην εργασία που ξεκινά τώρα γι' αυτό το ιδέασμα για την κινητικότητα. Είδατε πόσα νομοθετικά κείμενα θα χρειαστεί να εξετάσουμε ταυτόχρονα η θέληση του Κοινοβουλίου είναι να ρυθμιστεί το πρόβλημα. Γιατί ακόμα και αν η Επιτροπή έχει κάνει προσπάθεια για αυτό το πακέτο κινητικότητα, εμεί θέλουμε νίκη. Και άρα να ρυθμιστεί το θέμα που θέτει πρόβλημα. Το είπε η συνάδελφος, το θέμα της μαζικής αύξησης των καταχρήσεων. Εσείς πολλές φορές ήσασταν και μάρτυρες, μας είπατε πώς ζουν ορισμένοι εργαζόμενοι Ε, υπό απαράδεκτες συνθήκες στην Ευρώπη και Έχουμε μια κοινή θέληση, ναι, να πούμε ότι πρέπει να σταματήσει η ε, κατάσταση αυτή, αλλά υπάρχει και μια πραγματική βούληση για υποχρετικούς και δεσμευτικούς ελέγχους με κάτι το οποίο όλοι συμμεριζόμαστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του στόματος του Πρόεδρου τους είπε ίση εργασία για, για ίσους μισθούς, ίση μισθή για ίση εργασία και θέλουμε πλέον να μην κλείνουμε σε με τα μάτια απέναντι στο τι συμβαίνει γιατί αν το πράξουμε αυτό θα αφήσουμε η πόρτα και το δρόμο ανοιχτά στους δημαγωγούς που θέλουν να καταστρέψουν το ευρωπαϊκό project. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα στην Επιτροπή Μεταφορών. Σας ευχαριστώ όλους. friends, uh, παρακαλώ. Ετοιμαστείτε παρακαλώ για την ψηφοφορία κύριε και κύριοι να πάρετε